Ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, σας προτείνω να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Είμαστε στο σημείο 17 της ημερήσιας διάταξης και με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω την κυρία Σωτηρούλα Χαραλάμπους, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δεδομένου το ότι είμαστε πια στην Κυπριακή ε, προεδρία θα προεδρεύσει ε, στο ΕΠΣΚΟ που είναι ένα συμβούλιο αναφοράς για μας για ένα, σε μια πολύ σημαντική χρονική στιγμή όταν βλέπουμε τα κείμενα ε, τα οποία επεξεργάζεται το συμβούλιο αυτό. Κυρία Υπουργέ, δεν ξέρω αν χρειάζεται να σας παρουσιάσω, απλώς να υπενθυμίσω ότι έχετε ένα ιστορικό, ένα background ε, σε ε, κοινωνικές και διοικητικές επιστήμες, ότι έχετε εργαστεί στην Πανκυπριακή Εργατική Ομοσπονδία σε πολλές θέσεις πριν γίνετε ε, γενική γραμματέας του οργανισμού αυτού. Στη συνέχεια ήσασταν μέλος ε, της Βουλής των Αντιπροσώπων με το ΑΚΕΛ και δύο φορές ε, έχετε εκλεγεί. Μάλιστα με το χαρτοφυλάκιο το οποίο έχετε σήμερα γιατί ήσασταν πρόεδρος της Επιτροπής ε, Ίσων Ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπως επίσης και της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Θα ήθελα να σας πω και πάλι ότι είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μας να σας καλωσορίζουμε εδώ σήμερα. Είναι κάτι που συνηθίζεται όπως γνωρίζετε, αλλά επειδή θέλουμε να έχουμε και πολύ καλές βάσεις συνεργασίας με τις ε, ε, προεδρίες, ε, όχι για να κάνουμε κανένας είδους εξέταση, απλώς θέλουμε να γνωρίσουμε τις προεδρίες, να γνωρίζουμε εσά εσάς καλύτερα, να γνωρίζετε και εσείς τους κοινωνικούς εταίρους. Ε, και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για μας να γνωρίζουμε τους συνομιλητές μας στην Κυπριακή Προεδρία. Θα ήθελα με αυτά τα λόγια να σας δώσω το λόγο. Θα το γνωρίζετε, αλλά ε, να σας πω και εγώ ότι η Επιτροπή μας έχει ήδη τοποθετηθεί για τον ε, Γενικό Κανονισμό για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όπως επίσης και για το πρόγραμμα ε, ε, κοινωνικής πρωτοβουλίας. Η συγκήτριά μας είναι εδώ, είναι η κυρία Στάινρουκ και επίσης ε, για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Οι εργασίες μας έχουν λιγότερο προχωρήσει, αλλά είναι ένα ζήτημα για το οποίο ενδιαφέρονται πάρα πολύ τα μέλη της Επιτροπής μας. Όταν βλέπω τα στοιχεία ε, που θα πρέπει να επεξεργαστείτε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Ε, κάτι μου λέει ότι κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων ε, γύρω από τις δημοσιονομικές προοπτικές θα πάρουν πολύ χρόνο. Θέλουμε στο πλαίσιο της δικής μας Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων να συζητήσουμε και άλλα θέματα τα οποία μας απασχολούν όλος ιδιαίτερος την έκθεση του Αλεξάνδρου Σέρκας θα ήθελα να αναφέρω όλος ιδιαίτερος που αφορά νομοθετική πρόταση στον τομέα της αναδιάρθρωσης. Δεν θα ήθελα να σας πω περισσότερα ε, ως εισαγωγικά σχόλια. Ούτως ή άλλως τα μέλη της Επιτροπής μας θα σας θέσουν ερωτήσεις, είμαι βέβαιη. Οπότε σας δίνω να κάνετε εισαγωγή στη συζήτηση αυτή επί τη βάση όσων αυτών που θέλετε να μας πείτε σε σχέση με τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές. Προερχόμενοι και εγώ από την οικογένεια των κοινοβουλευτικών, γνωρίζω και αναγνωρίζω τον τεράστιο ρόλο που οι βουλευτές τόσο στο εθνικό αλλά και στο ευρωπαϊκό επίπεδο διαδραματίζουν στην ε, προσπάθεια για να υπάρξουν οι κοινέ συνισταμένες και εκείνες οι συγκλήσεις που θα βοηθήσουν τόσο στο εθνικό αλλά και στο πανευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα μέσα σε αυτές τις ε, δύσκολες ε, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, για να έχουμε εκείνες τις πολιτικές που θα μας επιτρέπουν να βγούμε από την κρίση και να δούμε τους πολίτες της Ευρώπης με αισιοδοξία στα μάτια και να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά. Γι' αυτό ε, θα ήθελα από την αρχή να πω ότι όχι απλά προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας, αλλά είμαι στην ε, διάθεσή σας ε, για ζητήματα που σας ενδιαφέρουν να προχωρήσουμε αυτή τη συνεργασία. Όπως έχω πει, η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την Ευρώπη είναι πολλέ οι πιέσει που αντιμετωπίζουν τα πλήστα κράτη-μέλη σε σχέση με την κοινωνική πολιτική και την πολιτική απασχόληση. Η κρίση έχει σημαντικές επιπτώσει στην ποιότητα ζωή των πολιτών. Οι ευάλωτε ομάδε του πληθυσμού διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Η ανεργία βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα. Ειδικότερα η ανεργία ανάμεσα στους νέους βρίσκεται σε πρωτοφανή επίπεδα και χρειάζεται να λάβουμε άμεσα μέτρα για να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Σε αυτό το πλαίσιο, το Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής καλείται να διαδραματίσει ένα συγκεκριμένο και δύσκολο ρόλο. Καλείται να διασφαλίσει ότι θα προχωρήσει με αποφασιστικότητα σε ανάπτυξη προσανατολισμένη στην απασχόληση με προσήλωση στο κοινωνικό πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους κοινωνικούς προσανατολισμούς της στρατηγικής Ευρώπη 2020, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την απασχόληση, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Όπως έχω ήδη πει, η Κυπριακή Προεδρία θεωρεί το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κομβικό στην ουσιαστική επίτευξη όλων όσων έχω προαναφέρει. Προσβλέπουμε στη στενή και επικοδομητική συνεργασία σας για την πρόθεση εκείνων των πολιτικών που θα βοηθήσουν την Ένωση μας να ανακάμψει σε συνθήκες ανάπτυξης και με κεντρικό στόχο την ευημερία και τη διασφάλιση υψηλού επίπεδου ποιότητας ζωής για κάθε πολίτη της Ένωσης. Από τον Νοέμβριο του 2012 έχουμε πραγματοποιήσει μια σειρά από επαφές με ευρωβουλευτέ μέλη των αρμόδιων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό είχα την χαρά και την τιμή να συναντηθώ με σας, κυρία Πρόεδρε, αλλά και με τους συντονιστές των ομάδων πολιτικών κομμάτων, καθές και συντονιστές συγκεκριμένων δοσιές. Οι συναντήσεις ήταν ιδιαίτερα επωφελείς, αφού είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για τις θέσεις του Κοινοβουλίου σε πολλά από τα θέματα που θα κληθούμε να χειριστούμε ως Προεδρία. Και περιμένουμε την επικείμενη επίσκεψη των μελών της Επιτροπής στο τέλος του Αυγούστου, που είμαι σίγουρη ότι θα είναι ακόμα μια εξαιρετική ευκαιρία για να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο σε θέματα που από κοινού θα μας απασχολήσουν το επόμενο εξάμεινο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του περασμένου Γενάρη σύστησε τη λήψη άμεσων και δραστικών μέτρων για αντιμετώπιση του πραγματικά πολύ σοβαρού προβλήματος της ανεργίας των νέων. Πριν από λίγες μέρες δε, υιοθέτησε το Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, το οποίο περιλαμβάνει τις δράσεις που στοχεύουν στην αναθέρμανση της ανάπτυξης, τις επενδύσεις και την απασχόληση. Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, χρειάζεται ταυτόχρονα με τη δημοσιονομική εξυγίανση να προωθούσουμε επενδύσεις για ανάπτυξη, που με τη σειρά τους θα ενισχύουν την απασχόληση και τη δημιουργία σταθερών και καλών θέσεων εργασίας. Η Κυπριακή Προεδρία έχει επιλέξει ως κεντρικό της μήνυμα το μήνυμα για μια καλύτερη Ευρώπη. Στόχος μας είναι να συνεισφέρουμε στην πρόθεση βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης που να βασίζεται στις αρχές της αλληλεγγύης με κύριο προσανατολισμό την παροχή ενός καλύτερου μέλλοντος για τις νεότερες γενιές. Μια από τις κύριες προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας είναι μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες. Προτεραιότητα κάτω από την οποία υπάγονται οι προτεραιότητες μας στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής. Να μου επιτρέψετε πολύ συνοπτικά να αναλύσω αυτές τις προτεραιότητες. Εστιάζονται στις ακόλουθες, στα ακόλουθα βασικά σημεία. Πρώτον, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής με έμφαση στην ευζοία των παιδιών. Η ευζοία των σημερινών παιδιών είναι αποφασιστικός παράγοντας για το μέλλον της Ευρώπης. Επενδύοντας στα παιδιά, επενδύουμε στην κοινωνική συνοχή αλλά και στην ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κυπριακή Προεδρία στοχεύει στην υιοθέτηση συμπερασμάτων τα οποία να εστιάζονται σε όλες τις πτυχές του θέματος της ευζοίας των παιδιών, της παιδικής φτώχειας και της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Πρόθεσή μας είναι όπως το κείμενο των συμπερασμάτων βασιστεί σε σχετική εργασία που ετοιμάζει η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας για τις κύριες αρχές και δείχτες που διέπουν την παιδική φτώχεια και ευζοία των παιδιών. Για το θέμα αυτό έχει προγραμματιστεί συνέδριο Προεδρίας τον Οκτώβριο του 2012, στο οποίο θα κληθεί να δώσει την δική του συνεισφορά και να συμμετάσχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η δεύτερη προτεραιότητα κάτω από την ευρύτερη προτεραιότητα για ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής σχετίζεται με το Ευρωπαϊκό Έτος για την ενεργό γύρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Στόχος της Προεδρίας είναι η οθέτηση διακήρυξης που θα σηματοδοτεί τη λήξη του έτους. Αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε ως Προεδρία στο πλαίσιο του έτους είναι ότι η ενεργός γύρανση δεν σημαίνει μόνο διατήρηση στην απασχόληση των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων, αλλά ενεργό συμμετοχή των μεγαλύτερων σε ηλικία πολιτών σε όλες τις διαστάσεις της κοινωνίας, καθώς και την ανάγκη για στήριξη της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Χρειαζόμαστε μια κοινωνία για όλους. Μια κοινωνία όπου η κάθε γενιά θα μπορεί να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες της και ταυτόχρονα μια κοινωνία όπου η μια γενιά θα μαθαίνει και θα παίρνει εμπειρίες από την άλλη. Η τελετή λήξη του Ευρωπαϊκού έτους θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2012 στην Κύπρο. Δεύτερη κυρία προτεραιότητα είναι η επένδυση σε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, νέες και αναβαθμισμένες δεξιότητες. Έμφαση θα δοθεί στην καταπολέμηση της ανεργίας ανάμεσα στους νέους, συνδέοντας αυτή την προτεραιότητα με την πρωτοβουλία της Επιτροπής Ευκαιρίες για τους Νέους, καθώς και με τα ζητήματα του πακέτου απασχόλησης που παρουσίασε η Επιτροπή τον Απρίλιο του 2012 και συνδέονται με την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Πρόθεση της Κυπριακής Προεδρίας είναι η έκδοση συμπερασμάτων για το θέμα αυτό, στα οποία θα περιλαμβάνονται ζητήματα που σχετίζονται με ευκαιρίες κατάρτισης, όπως είναι τα συστήματα μαθητείας και τα συστήματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, οι εργασιακές συνθήκες των νέων και η σύζευξη των προσόντων και προσδοκιών των νέων με τις ανάγκες της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Για το θέμα αυτό θα πραγματοποιηθεί συνέδριο Προεδρίας για την νεανική απασχόληση τον Οκτώβριο του 2012 στην Κύπρο. Τρίτη προτεραιότητα είναι η ενδυνάμωση των συμμετοχικών διαδικασιών και της εμπλοκής των κοινωνικών εταίρων των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των τοπικών αρχών στην υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 σε ό,τι αφορά ειδικά τους στόχους της απασχόλησης και της φτώχειας. Η επιτυχής υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 εξαρτάται από τη συμμετοχή όλων των τμήματων της κοινωνίας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο για να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής Ευρώπη 2020, μαζί με τις κυβερνήσεις χρειάζονται να δραστηριοποιηθούν όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Κοινωνική εταίροι, ΜΚΟ, τοπικές αρχές. Έχουν σημαντικό και βασικό ρόλο τόσο στη διαμόρφωση των πολιτικών, όσο και στη διαδικασία υλοποίησης των πολιτικών. Σε αυτό το σημαντικό θέμα, η Κυπριακή Προεδρία αποφάσισε να αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της άτυπης συνάντησης Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο τις αμέσως επόμενες μέρες, τις 12 και 13 του Ιούλη και στην οποία έχει προσκληθεί να συμμετάσχει και η Επιτροπή σας και με χαρά πληροφορούμε ότι θα είναι μαζί μας η αγαπητή κυρία Πρόεδρος της Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά στα συγκεκριμένα ντοσιέρ που θα τύχουν χειρισμού στο Συμβούλιο μας, Γνωρίζετε ότι υπάρχουν πολλά έκρημη θέματα, ήδη έχετε θίξει στην εισαγωγή σας κάποια από αυτά και πρόσθετα αναμένεται ένας σημαντικός αριθμός νέων πρωτοβουλειών εντός του 2012. Ξέρουμε ότι μας περιμένει πολλή δουλειά και ότι αρκετά από τα θέματα που καλέμαστε να χειριστούμε είναι πολύπλοκα. Θα επιδιώξουμε να πετύχουμε ουσιαστική πρόοδο στην πρόθεση των σημαντικότερων νομοθετικών πρωτοβουλειών με πνεύμα διαλόγου και συνένεσης, ενεργώντας ως έντιμοι διαμεσολαβητές τόσο εντός του Συμβουλίου όσο και μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μεταξύ των νομοθετικών πρωτοβουλειών στις οποίες η Κυπριακή Προεδρία θα δώσει προτεραιότητα είναι η οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων. Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών για τις διασυναριακές δραστηριότητες των επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά μπορεί να προωθηθεί μέσω της παροχής υψηλού επίπεδου προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Θεωρούμε ότι η πρόταση οδηγίας θα βοηθήσει στην καλύτερη εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για προστασία των αποσπόμενων εργαζομένων και θα συνεισφέρει σημαντικά στην αποτροπή φαινομένων εκμετάλλευσης εργαζομένων. Είναι πιστεύω κοινός στόχος όλων μας να εργαστούμε προς τη βελτίωση της κινητικότητας των εργαζομένων με τρόπο που να γίνονται σεβαστές οι αρχές της ελεύθερης διακίνησης και της διαφύλαξης αξιοπρεπώς συνθηκών εργασίας και να μην δημιουργούνται φαινόμενα κακών εργασιακών συνθηκών και του ανταγωνισμού. Σε ό,τι αφορά στον κανονισμό για το δικαίωμα σε συλλογική δράση, αφού έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία της κίτρινης κάρτας, θα αναμένουμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως στο κατά πόσο προτίθεται να διατηρήσει, τροποποιήσει ή αποσύρει την πρόταση. Τα θέματα ασφάλειας και υγείας είναι ψηλά στην ατζέντα της Κυπριακής Προεδρίας. Επομένως, η οδηγία για προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που προέρχονται από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι ακόμα μια νομοθετική πρόταση στην οποία θα δώσουμε προτεραιότητα. Είναι βέβαια ένα δύσκολο και τεχνικό θέμα, αλλά παράλληλα έχει και ένα απλό και συγκεκριμένο στόχο, την παροχή επαρκούς προστασίας των εργαζομένων. Με γνώμονα αυτή την αρχή σκοπεύουμε να εργαστούμε εντατικά για την εξέβρεση κοινού εδάφους για την επίτευξη συμφωνίας η οποία να διασφαλίζει επαρκώς την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Η Πολωνική και η Δανική Προεδρία έχουν εργαστεί εντατικά σε σχέση με την πρόταση αυτή και θα ήθελα ιδιαίτερα να τους ευχαριστήσω. Επί Δανικής Προεδρίας έχει επιτευχθεί καταρχή συμφωνία στο Συμβούλιο αναφορικά με τα παραρτήματα της οδηγίας τα οποία αφορούν στο είδος, αριθμός, αριθμό και ύψος των οριακών τιμών έκθεσης και των τιμών ανάληψης δράσης και η δική μας Προεδρία θα συνεχίσει την εργασία από εκεί που έχει μείνει έχοντας επίγνωση και τους χρονικούς περιορισμούς που επιβάλλουν την επίτευξη συμφωνίας το συντομότερο δυνατό. Στόχος μας είναι να υπάρξει γενική προσέγγιση στο Συμβούλιο του Οκτώβρη. Εκείνο που αναμένουμε λαμβάνοντας υπόψη και το επίγον του θέματος είναι τη συνεργασία σας για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε τελικό αποτέλεσμα. Με την ευκαιρία θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η Κυπριακή Προεδρία προγραμματίζει συνέδριο στην Κύπρο σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία με θέμα «Εργαζόμαστε μαζί για το μέλλον της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στην Ευρώπη». Σε ό,τι αφορά τις δύο προτάσεις που συνδέονται με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ο κανονισμός για το πρόγραμμα κοινωνικής αλλαγής και καινοτομίας, πιστεύουμε ότι έχει πολύ βασικό ρόλο να επιτελέσει στην παροχή οικονομικής στήριξης για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την προώθηση ψηλού επίπεδου απασχόλησης, τη διασφάλιση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και την βελτίωση των εργασιακών συνθήκων. Όσο εκ τούτου είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας με στόχο την επίτευξη συμφωνία στο θέμα. Ως προς τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, αναμένουμε δύσκολες διαπραγματεύσεις. Οι αλλαγές που παρατηρούνται στο παγκόσμιο εμπόριο όμως δεν είναι ένα βραχυπρόθεσμο φαινόμενο. Είναι μια μόνιμη κατάσταση η οποία θα εντείνεται με το καιρό. Το Ταμείο έχει ουσιαστική συνεισφορά στη στήριξη των εργαζομένων που έχουν χάσει τη δουλειά τους λόγω της παγκοσμιοποίησης. Για το σκοπό αυτό θα εργαστούμε με στόχο την εξέβρεση κοινών συνισταμένων για την περαιτέρω πρόθεση του θέματος. Και για τα δύο θέματα έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχουμε ενημερωθεί για τους προβληματισμούς σας. Η Προεδρία, σε ένα πνεύμα ειλικρινούς διαλόγου, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να μεταφέρει τις θέσεις σας στο Συμβούλιο με στόχο την εξέβρεση ισορροπημένων κοινά αποδεκτών λύσεων. Σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θέλω να τονίσω ότι η Κυπριακή Προεδρία θεωρεί ότι το Ταμείο παραμένει ένα βασικό εργαλείο για τη στήριξη των πολιτικών για ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, με σεβασμό στις εθνικές αρμοδιότητες των κρατών μελών ή περιφερειών. Ειδικότερα τώρα, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για την Ένωση. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι ακόμη πιο σημαντικός, καθώς στηρίζει ενεργά την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Το Ταμείο έχει πρωταρχικό ρόλο να διαδραματίσει στην υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και επιθυμούμε να αναδείξουμε αυτό το ρόλο του Ταμείου ως εργαλείο κοινωνικής επένδυσης και υλοποίησης της στρατηγικής. Χαιρετίζουμε την εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον κανονισμό που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου, αλλά και στην πολιτική συνοχή και προσβλέπουμε και σε αυτό το κεφάλαιο στη συνεργασία σα. Η Κυπριακή Προεδρία θα συνεχίσει την εργασία σε σχέση με τις προτάσεις αποφάσεων του Συμβουλίου για λήψη εντολής διαπραγμάτευσης με τα αντίστοιχα Συμβούλια Σύνδεσης αναφορικά με τις συμφωνίες σύνδεσης για θέματα κοινωνική ασφάλισης με την Αλβανία, το Μαυροβούνιο, το Σαν Μαρίνο και την Τουρκία. Επίσης, προτιθέμεθα να καταβάλουμε προσπάθεια ώστε να αρχίσουν ξανά οι συζητήσεις στο Συμβούλιο αναφορικά με την οδηγία για τα συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο το σύμφωνο της ενιαίας αγοράς, όσο και συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κάνουν αναφορά στο θέμα αυτό επισημένοντας την ανάγκη ενίσχυσης της απόκτησης και διατήρησης των συνταξιοδοτικών και άλλων δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων. Πρόσθετα θα συνεχίσουμε την εργασία σε σχέση με την ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση, συνεχίζοντας τη βάση της εργασίας που έκαναν η Πολωνική και η Ιδανική Προεδρία σε σχέση με τις πρόνοιες που αφορούν την ηλικία ως παράγοντα διάκρισης, αφού είναι η γενική διαπίστωση του Συμβουλίου ότι εν λόγω πρόνοιες χρήζουν περαιτέρω εξέτασης. Μια σημαντική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα της ισότητας και η οποία συνδέεται άμεσα με την απασχόληση σχετίζεται με το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Έχουμε και μια ιδιαίτερη εθνική ευαισθησία σε αυτό το θέμα, αφού η Κύπρος συγκαταλέγεται στα κράτη-μέλη με υψηλό χάσμα αμοιβών, παρά την πρόοδο που σημειώνεται τα τελευταία χρόνια στη μείωση του χάσματος αμοιβών, που είναι αυτή τη στιγμή γύρω στο 21%. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι αιτίε του χάσματος είναι πάρα πολλέ και ότι χρειάζεται να εργαστούμε σε πολλαπλά επίπεδα, τόσο στο επίπεδο των μισθολογικών κλιμάκων, αλλά και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το εκπαιδευτικό σύστημα, με τις πολιτικές απασχόλησεις, για να μπορέσουμε να έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να σας ενημερώσω ότι κάτω από την αιγίδα της Προεδρίας θα πραγματοποιήσουμε συνέδριο με τη συμμετοχή κυβερνήσεων, συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων για το χάσμα των αμοιβών τον Οκτώβριο του 2012. Σε αυτό το συνέδριο οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τις διάφορες προκλήσεις αλλά και να προσδιορίσουν καλές πρακτικές. Ένας από τους στόχους του συνεδρίου είναι να αναδειχθούν πρακτικές και μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν στο επίπεδο των επιχειρήσεων προκειμένου να εξαλειφθεί το χάσμα των αμοιβών. Για τη θεματολογία του συνεδρίου έχουμε μελετήσει και αξιοποιήσει την πραγματικά αξιόλογη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με τις συστάσεις προς την Επιτροπή για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβή. Θα κλείσω την ενημέρωσή μου με ορισμένα από τα σημαντικότερα συνέδρια που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας στα θέματα κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής απασχόλησης πέραν των όσων έχω ήδη αναφέρει. Τον Δεκέμβριο του 2012, 5 με 7 του Δεκέμβρη, θα πραγματοποιηθεί στι Βρυξέλλες η ετήσια σύνοδο τη Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Θα πραγματοποιηθεί επίση η Υπουργική Σύνοδο των Υπουργών Εργασία και Απασχόληση Ασία και Ευρώπη στι 25 με 26 Οκτωβρίου 2012 στο Βιετνάμ, καθώ και η Υπουργική Διάσκεψη για την Τρίτη Ηλικία που διοργανώνεται από την UNESCO και το ε, Αυστριακό Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Προστασίας των Καταναλωτών στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2012 στη Βιέννη, ένα συνέδριο το οποίο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία και ενδιαφέρον λόγω του φετινού Ευρωπαϊκού Έτους. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ευρωβουλευτές, για ακόμα μια φορά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και είμαι στη διάθεσή σας για τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς οι δύο συντονιστές, ο κύριος Τσαμπαόρη, ο ο κύριος Ορύπρωτα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω την Υπουργό Χαίρομαι πολύ που υπάρχει ιδιαίτερη, ε, ιδιαίτερα ε, κοινοβουλευτικός φιλική διάθεση από την πλευρά σας ε, και βλέπω ότι η Κυπριακή Προεδρία ε, επιθυμεί συνεργασία με την Επιτροπή μας. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα πράγματα που αναφέρατε και εσείς και έχω και μερικές ερωτήσεις. Στο ΕΛΚ πιστεύουμε ότι η σημαντικότερη προτεραιότητα είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Υπάρχει όμως το εξής δίλημα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη κάποιες κοινωνικές αξίες. Από την άλλη όμως, πρέπει να υπάρξουν και οι απαραίτητες προϋποθέσεις και η ευελιξία, ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει η οικονομία νέες θέσεις απασχόλησης. Συνεπώς, τα κοινωνικά ζητήματα βρίσκονται στο περιθώριο και το πρώτο μου ερώτημα συνεπώς είναι το εξής. Σε σχέση με τη δέσμη μέτρων για την απασχόληση, σε ποιους τομείς θεωρείτε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε για να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μειώσουν το διοικητικό τους ε, φόρτο, τη μείωση των φόρων. Κάποια τέτοια ζητήματα σίγουρα θα συζητηθούν. Εμείς ε, ως μέλη του ΕΛΚ δεν θέλουμε κάτι το καινοφανέ ε, σε σχέση με την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων. Θεωρούμε ότι είναι μια καλή οδηγία. Βεβαίω, υπάρχουν κάποια προβλήματα στην πράξη. Θα έχετε ακούσει βεβαίω ότι εκ μέρου του ΕΛΚ έχουμε ενημερώσει, Επίτροπο, ότι το υπόλοιπο τμήμα της δέσμης, ε, η πρόταση Μόντι δύο και μετά τη χρήση της κίτρινης κάρτας ε, θεωρούμε ότι δεν έχει κανένα νόημα. Πιστεύουμε ότι πρέπει να αποσυρθεί η πρόταση. Δεν θεωρούμε ότι αξίζει τον κόπο να ξοδέψουμε ενέργεια για πράγματα τα οποία δεν χρήζουν καμίας υποστήριξης. Για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι εδώ δίπλα μου η συγχύτρια, ούτως ή άλλως ε, θα το αναφέρει και εκείνη. Έχω κάποιες επιφυλάξεις. Είναι ένα πολύ τεχνικό ζήτημα. μένονται οι εντονότερες ε, ε, πολιτικές συζητήσεις πίσω από κάτι που φαινομενικά είναι απλώς ε, ένα τεχνικό πρόβλημα. Οπότε ελπίζουμε συνεργασία με τους κοιόδης συζητητές και με τους συναδέλφους ευρωβουλευτές. Ελπίζουμε στο Κοινοβούλιο να λυθεί το θέμα. Είμαι, ε, καταλαβαίνω βέβαια ότι εσείς στο Συμβούλιο έχετε μικρότερο περιθώριο ελιγμών. Ευχαριστούμε για τον κατάλογο των ε, διασκέψεων. Θα προσπαθήσουμε να παραστούμε σε όσες περισσότερες μπορούμε. Επίσης, ε, τη δήλωσή σας για την ενεργό γύρανση τη θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική. Υπήρξαν πολλές ε, Πρωτοβουλίε ε, από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επεξεργαζόμαστε και άλλες. Πιστεύω ότι θα είναι καλή η συνεργασία μας και θα ήθελα να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία για τους επόμενους έξι μήνε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σέρκας. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να καλωσορίσω πρώτα απ' όλα την κυρία Υπουργό στην Επιτροπή μας. Και Ίσως να ζητήσω και συγγνώμη για ένα ραντεβού που αναγκαστήκαμε να ακυρώσουμε στην ε, Κύπρο, αλλά τελικά νομίζουμε ότι έχει αναβληθεί για τον Αύγουστο, αν κατάλαβα καλά, οπότε εκεί θα έχουμε την χαρά να ανταλλάξουμε απόψεις. Τώρα επιτρέψτε μου να κάνω μια γενική εκτίμηση ε, της παρουσίας που κάνετε και μετά να κάνω κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα. Η γενική αποτίμηση, αν θέλετε, που μπορώ να κάνω, έχει να κάνει εξή. Οι επαφέ που είχαμε και με την Προεδρία στην προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο μα επέτρεψαν να τοποθετήσουμε αυτή τη συζήτηση στην ευρύτερη ευρωπαϊκή ιστορία. Άρα, δηλαδή, πώ η Προεδρία εντάσσεται α, σε αυτή την ιστορία. Αυτό το εξάμεινο δεν θα είναι μόνο ιστορικό, πιστεύω, μόνο για εσά, γιατί για πρώτη φορά αναλαμβάνετε την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γιατί ζούμε μια ιστορική στιγμή στην Ευρώπη. Είναι στιγμές που επιταχύνεται η ιστορία και νιώθω ότι ζούμε μια τέτοια ιστορική στιγμή. Κύριε Υπουργέ, η Ευρώπη, η κοινωνική, πώς κινείται παράλληλα με την ε, Ευρωζώνη, με το νέο νόμισμα. Και θέτει ένα ερώτημα, αν θέλετε αυτό. Ή θα προχωρήσουμε σε βαθύτερη ένωση ή θα διαλυθούμε. Υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να τα επιλύσουμε. Δεν αρκούν οι μη για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Χρειάζεται λοιπόν ένας οδικός χάρτης, ένα roadmap για να μα οδηγεί στην έξοδο από την κρίση. Δηλαδή χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια πολιτική διευθέτηση κατάσταση. Η διευθέτηση απλά μα οδηγεί μαθηματικά στην καταστροφή και στην ε, πλήρη απελπισία για τους Ευρωπαίους πολίτες. Οι πολίτες θέλουν ανάπτυξη, θέλουν απασχόληση και θέλουν να διατηρήσουν το επίπεδο ε, το βιωτικό τους. Εσείς λοιπόν έχετε αντιμετωπίσει μια σημαντικότερες πολιτικές απασχολεί τους πολίτες. Ήδη στο Συμβούλιο ακούγονται διάφορες φήμες ότι μπορούμε να κινηθούμε σε μια νέα πολιτική, ότι μπορούμε να αλλάξουμε σελίδα, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη ώστε να εμπνεύσουμε ελπίδα στους πολίτες μας. Αυτά γενικά κύριε Υπουργέ. Εδώ θέλω να πω ότι στην, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθούμε η Επιτροπή Απασχόλησης να έχει εξίσου ισχυρή φωνή όπως ε, η Επιτροπή Οικονομικών. Ρωτώ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι επίτροποι που έχουν ε, τα αρμόδια χαρτοφυλάκια, τα οικονομικά δηλαδή και την απασχόληση. Θέλω να σας καλέσω στις επαφές μαζί τους να δώσετε μάχη, κύριε Υπουργέ. Δεν μπορεί το ΕΚΟΦΗ να είναι το μόνο συμβούλιο που ακούγεται σε όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει και το δικό σας συμβούλιο, το ΕΠΣΚΟ, είναι ένα συμβούλιο που θα πρέπει να ακουστεί πολύ ισχυρά η φωνή του σε όλη την Ευρώπη. Και τώρα να θέσω κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα. Είπατε κύριε Υπουργέ ότι το θέμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ε, είναι μια περίπλοκη ιστορία. Κοιτάξτε, είναι από τα λίγα επιτεύγματα της Ευρώπης έναντι εκατοντάδων χιλιάδων εργαζόμενων που αντιμετωπίζουν το θέμα της ανεργίας ε, λόγω της μετεγκατάστασης ε, επιχειρήσεων. Αν λοιπόν δεν επιτύχουμε σε αυτό μας το στόχο, θα κάνουμε δυστυχώς ένα τεράστιο βήμα πίσω σε σχέση με τα επιτεύγματα. Ξέρετε, είναι ευκολή η καταστροφή σήμερα. Υπάρχουν μέλη στο Συμβούλιο που θέλουν να αν θέλετε, να νοθεύσουν αυτή την ε, ισχύ και τη δυναμική που μπορούμε να έχουμε, προσπαθώντας να μοιράσουν κονδύλια αλλού. Κοιτάξτε, δεν πιστεύω ότι η λύση ε, είναι να θυσιάσουμε κάποια μερίδα πολιτών και εργαζομένων για να υπερασπιστούμε άλλους όπως τους αγρότες, την πολιτική γεωργίας κτλ είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και θέλω να πω ότι η κοινωνική πολιτική είναι ένα σύμβολο για την Ευρώπη και δεν μπορούμε να την καταστρέψουμε. Είναι ένα σύμβολο επίσης των, των Ευρωπαϊκών Συμβασμών έναντι των Ευρωπαίων εργαζομένων που είναι τα θύματα των αντικαταστάσεων των επιχειρήσεων. Κάτι άλλο. Για το θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα ε, είναι οι νέες προτάσεις του νέου πακέτου για την απασχόληση και θέλουμε τη δική σας βοήθεια. Και τέλος, ε, κύριε Υπουργέ, είπατε ότι θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη δικαιοσύνη στα θέματα των εργαζομένων. Όσον αφορά την απόσπαση των εργαζομένων, ξέρετε, ακούσαμε τη θέση του εκπροσώπου του ΕΛΚ. Εμείς, που σοσιαλιστές, θέλουμε μια άλλη πολιτική. Θέλουμε αλλαγή τη πολιτική. Θεωρούμε ότι είναι μια πολύ κακή οδηγία. Έχουμε την ομολογία του ΔΕΚ και ήδη δημιουργούνται τεράστιε συγκρούσει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα ερμηνεία οδηγία και τι ζητούμε κάτι απλό. Θα πρέπει οι εργαζόμενοι που έχουν τη θέση εργασία και παρέχουν τι υπηρεσίε να λαμβάνουν τι ίδιε απολαυέ δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται οι μετανάστες ως μία δύναμη εργατικού δυναμικού χαμηλού κόστους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, θα ήθελα να σας δώσω το λόγο να απαντήσετε σε αυτές τις δύο ερωτήσεις. Ε, ίσως λίγο πιο σύντομα από το χρόνο που πήραν οι συνάδελφοι να σας τις θέσουν, γιατί οχτώ ακόμη ομιλητές θέλουν να λάβουν το λόγο. Έχετε το λόγο. για να απαντήσετε στους δύο συντονιστές μας του ΕΛΚ και των Σοσιαλιστών. Θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ στην ε, παράκλησή σας. Ε, και για να ανταποκριθώ θα προσπαθήσω μέσα από τις δύο τοποθετήσεις και τα ερωτήματα να αναδείξω ε, εκείνα τα ζητήματα που νομίζω ότι είναι σημαντικά. Και το σημαντικότερο νομίζω που αναδεικνύεται από τις συζητήσεις και εδώ και καθημερινά είναι ότι έχουμε περάσει και περνούμε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο στην Ευρώπη σχεδόν σε όλες ε, τις ε, χώρες ε, οι κυβερνήσεις αλλά και οι λαοί μας έχουν περάσει μέσα από δύσκολες πολιτικές για να καταφέρουμε να πετύχουμε δημοσιονομική εξυγίανση. Βιώνουμε πάρα πολύ ψηλά ποσοστά ανεργίας, αυτό αφορά και τη δική μου χώρα. Και είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυναμική η οποία αυτή τη στιγμή δημιουργείται μέσα από διάφορες πρωτοβουλίες και πολιτικές. Ειδικότερα θα ήθελα να αναφερθώ στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Σύμφωνο για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη και να κάνουμε το μεγάλο αναγκαίο βήμα. Και το μεγάλο αναγκαίο βήμα το οποίο έχουμε όλοι ανάγκη αυτή τη στιγμή είναι πώς κατευθύνουμε τις πολιτικές μας και τους πόρους μας χωρίς να εγκαταλείπουμε την ανάγκη να έχουμε υγιείς ε, προϋπολογισμούς, αλλά να αξιοποιήσουμε αυτούς τους προϋπολογισμούς για την ανάπτυξη και για την δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό ισχύει και για το εθνικό επίπεδο, αυτό ισχύει και για το ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάτω από το ίδιο πρίσμα, ως Προεδρία, βλέπουμε την αξιοποίηση και διαφόρων άλλων πρωτοβουλειών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα το πακέτο απασχόλησης και την πρωτοβουλία για τους νέους. Η κάθε χώρα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και δεν μπορούμε να βάλουμε όλες τις χώρες κάτω από το ίδιο πλαίσιο και κάτω από τις, ε, ε, ίδιες κατευθύνσεις. Εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία είναι να βρούμε την αναγκαία ισορροπία από τη μια σε πολιτικές που θα δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δημιουργούν θέσεις εργασίας, αλλά ταυτόχρονα σε αυτή τη διαδικασία να μην υποβιβάζεται και να μην αφήνεται σε δεύτερη μοίρα η ποιότητα της εργασίας και βασικά εγώ θα έλεγα όχι εργατικά δικαιώματα, αλλά ανθρώπινα δικαιώματα, για τα οποία η Ευρώπη πρέπει να είναι περήφανη, γιατί είναι αυτή που έκτισε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Άρα εγώ σχολιάζοντας ε, ε, τα, ερωτήματα, τα σχόλια καλύτερα και των δύο συντονιστών, θα έλεγα ότι η Κυπριακή Προεδρία, αξιοποιώντας ακριβώς αυτή τη δυναμική που έχει ε, δημιουργηθεί αυτή τη ε, στιγμή θα προσπαθήσει μέσα από τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει να γίνουμε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι προς ε, αυτή την, κατεύθυνση. Ακριβώς γι' αυτό γιατί έχω πει προηγουμένως ότι δεν μπορούμε να έχουμε συνταγές που να ανταποκρίνονται σε όλους. Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, η μείωση της φορολογίας της εργασίας σε κάποιες χώρες που είναι ιδιαίτερα ψηλή μπορεί να είναι μια θετική πολιτική προς την κατεύθυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας αλλά αυτό πρέπει να το κοιτάζουμε πάντοτε μέσα στο πλαίσιο το οποίο έχω ε, πει προηγουμένως. Για την απόσπαση των ε, εργαζομένων και για τον ε, κανονισμό Μοντιδίου. Εμείς εκκινούμε από μια θέση οποία, η οποία πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι η κοινή συνισταμένη ότι είμαστε μια Ευρώπη των 27, μια Ευρώπη η οποία πρέπει στην πράξη να ενθαρρύνει την κινητικότητα μεταξύ των εργαζομένων, να δίνει δυνατότητες στους Ευρωπαίους πολίτες να μπορούν να εργάζονται σε ε, οποιαδήποτε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα όμως, την ίδια ώρα, σημείο εκκίνησης είναι ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνεται κάτω από πλαίσια που να διασφαλίζουν την ισότητα της μεταχείρισης, να αποτρέπουν την κακή χρήση της διακίνησης των, ε, των εργαζομένων, να διασφαλίζουν, την, όπως έχω πει, την ισότητα μεταξύ των εργαζομένων. Κάτω από αυτό το πλαίσιο προσεγγίζουμε και την εφαρμοστική οδηγία θα εργαστούμε στο πλαίσιο του Συμβουλίου για να προχωρήσουμε τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει επί Δανικής Προεδρίας. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά θεωρούμε ότι υπάρχουν στοιχεία πάνω στα οποία μπορούμε να εργαστούμε στο πλαίσιο του Συμβουλίου για να χτίσουμε και να δώσουμε ε, αυτό το οποίο έχει ανάγκη σήμερα η Ευρώπη στα πλαίσια της διασφάλισης της έννοιας, της κινητικότητας αλλά ταυτόχρονα και των ε, δικαιωμάτων των εργαζομένων. Σε ό,τι αφορά ε, το Μοντιδίο, σαφέστατα η κίτρινη, κάρτα, η κίτρινη κάρτα που έχει δοθεί από εθνικά κοινοβούλια έχει δημιουργήσει μια καινούργια κατάσταση δεν μπορούμε παρά να αναμένουμε ποια θα είναι η θέση της Επιτροπής και σαφέστατα και οι ανησυχίες και οι απόψεις οι οποίες έχετε εκφράσει εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικές στο να αντιληφθούμε και εμείς ως Προεδρία τις ευαισθησίες που υπάρχουν και στο Ευρωκοινοβούλιο ε, και, ε, και σε, στα Εθνικά Κοινοβούλια γύρω από αυτό το θέμα. Ένα σχόλιο αναφορικά με το ρόλο του Συμβουλίου ΕΠΣΚΟ ε, ε, στην, όλη διαδικασία ε, των, πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να υπογραμμίσω ότι συμμετέχοντας στο Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής σχεδόν για πέντε χρόνια τώρα, αυτά είναι ένα, είναι ένα από τα ζητήματα που μαζί με όλους τους συναδέλφους Υπουργούς Απασχόλησης έχουμε πάρα πολλές φορές συζητήσει. Αυτό είναι και ο λόγος πρέπει να πω που έχουμε αποφασίσει ένα, μία από τις συζητήσεις που θα κάνουμε στο πλαίσιο του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης στην Κύπρο να διασυνδεθεί με το ρόλο του Συμβουλίου αλλά και των άλλων παιχτών, όπως έχω πει των κοινωνικών εταίρων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων ε, και των ε, τοπικών αρχών στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Διότι πιστεύουμε ότι η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου πρέπει να είναι μια διαδικασία όπου το κάθε Συμβούλιο να νιώθει ότι έχει συμμετοχή και ρόλο μέχρι την, ε, τελική φάση. Δεν θα ήθελα να υποσχεθώ μεγάλα λόγια. Εκείνο το οποίο θέλω να υποσχεθώ ότι θα προσπαθήσουμε σε αυτό το εξάμεινο αυτή την ε, βασική έννοια και αρχή να την διαπεράσουμε στον τρόπο με τον οποίο η Κυπριακή Προεδρία θα ασκήσει τον ε, δικό της ρόλο και είμαι σίγουρη ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα έχουμε και την συνεργασία των, ε, των άλλων μου συναδέλφων. Ε, έχω την εντύπωση, κυρία Πρόεδρε, ότι έχω σχολιάσει τις ε, πρώτες ε, τοποθετήσεις που έχουν γίνει από τους κυρίους ευρωβουλευτές. Yeah. Alors, on va faire... Μάλιστα. Η κυρία Στάινρουκ και ο κύριος Πουπάκης μετά. Η κυρία Στάινρουκ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, Τις ε, προηγούμενες εβδομάδες μας προσφέρθηκε η ευκαιρία, ε, λόγω και της έκθεσης ε, την οποία επεξεργάζομαι εγώ, να ανταλλάξουμε απόψεις. Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία να συζητήσουμε, αλλά οι σημερινές μου ερωτήσεις αφορούν την καινοτομία και την κοινωνική αλλαγή, κάτι το οποίο θεωρεί σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το αποκαλεί καινοτομία για την απασχόληση. Γνωρίζετε λοιπόν ότι η δική μας η Επιτροπή ε, αποφάσισε με πλειοψηφία. Σήμερα μάλιστα είχαμε την ε, σύμφωνη γνώμη σχεδόν όλων των συναδέλφων. Ελάχιστοι διαφώνησαν. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι στο πρόγραμμα αυτό πρέπει να παρισφρήσει ένας περαιτέρω άξονας που αφορά στην αντιμετώπιση αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Γίνονται πάρα πολλές κουβέντες, πολλά λέγονται, αλλά κατά τη δική μας άποψη υπάρχει η ευκαιρία να αναλυφθούν πρωτοβουλίες, να δρομολογηθούν συγκεκριμένα προγράμματα. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που η Κυπριακή Προεδρία θεωρεί ως μία από τις βασικές της προτεραιότητες την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Γι' αυτό λοιπόν ε, παρακαλώ για την υποστήριξή σας και στο θέμα αυτό, διότι ο τομέας αυτός, στον τομέα αυτό μπορούμε να προχωρήσουμε μόνο εφόσον συμφωνήσουμε ότι χρειαζόμαστε επιπρόσθετα κονδύλια. Εμένα λοιπόν με ενδιαφέρει το πώς αξιολογείτε εσείς αυτή την πρωτοβουλία και πώς θεωρείτε ότι θα την εξολογήσουν και οι συνάδελφοί σας στο Συμβούλιο. Αυτή είναι η μία μου παράκληση. Και τώρα το δεύτερο σκέλος της ερώτησής μου αφορά το εξής. Αφορά το πρόγραμμα OIRES. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει από το 2014 οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές τα προβλήματα αυτών των εργαζομένων να επιληθούν στο πλαίσιο του μηχανισμού που υφίσταται. Γιατί αποδείχθηκε ότι μέχρι τώρα υπάρχει πρόβλημα κινητικότητας των εργαζομένων ε, στις παραμεθόριες περιοχές. Όμως, και εσείς το είπατε, είναι απαραίτητο να βελτιώσουμε την κινητικότητα των εργαζομένων. Πρέπει να αρθούν τα μειονεκτήματα που υφίστανται. Εχθές ε, ήμουνα στο εργοστάσιο της ε, Mercedes, ιδίω των φορτηγών, τους επισκέπτηκα επιτόπου και μου είπαν ότι τα πράγματα είναι τραγικά. Δηλαδή υπάρχουν εργαζόμενοι σε παραμεθόριες περιοχές και εγώ έρχομαι από μια τέτοια παραμεθόρια περιοχή. Αυτοί λοιπόν χρειάζονται περισσότερες ε, συμβουλές, ε, συστάσεις. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να γίνεται εξοικονόμηση κονδυλίων όσον αφορά την παροχή συμβουλών σε αυτούς τους εργαζόμενους. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας παρακαλέσω αυτό το θέμα να το ενστερνιστείτε. Η δική ε, Επιτροπή Επιτροπή έχει διαπιστώσει ότι μπορούν να παραμείνουν οι αδελφοποιήσεις παραμεθόρων περιοχών στο πρόγραμμα ΟΙΡΕΣ. Για να το κάνουμε όμως αυτό χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω από του συναδέλφου να είναι λίγο πιο σύντομοι. Κυρία Στάνιρουκ, δεν σα διέκοψα, αλλά κακώ. Κύριε Πουπάκη. Και μετά, ο κύριο Κρίστενσεν, ο κύριο Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Υπουργέ. Η ανάληψη τη Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την Κύπρο πραγματοποιείται, όπω και εσεί είπατε, σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη συγκυρία για την προοπτική τη Ευρωπαϊκή Οικονομία, αλλά και για τη συνοχή τη Ευρωπαϊκή κοινωνία. Μπορεί οι αποφάσει τη τελευταία Συνόδου Κορυφή να είναι ενθαρρυντικέ για μια ουσιαστική κοινωνική και παραγωγική ανάκαμψη, όμω υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που απαιτούν άμεση λύση, όπω είναι η ανεργία, η καταπολέμηση του φαινόμενου τη φτώχεια, η ενίσχυση τη ποιοτική απασχόληση και η προάσπιση τη ασφάλεια στην εργασία. Και αυτό το λέω έχοντα παράδειγμα τη χώρα μου, όταν ένα στου δύο νέου, και επειδή μιλάμε για του νέου, είναι εκτός αγοράς εργασίας, ενώ το 68% του πληθυσμού ζει στο όριο της φτώχειας, με τους αστέγους να πολλαπλασιάζονται, τις αυτοκτονίες λόγω ανέχειας να αποτελούν μια τραγική καθημερινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα ήθελα να μάθω πώς η Κυπριακή Προεδρία σκοπεύει να προωθήσει ένα ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο για αυτά τα ζητήματα, ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει να αναλάβει για αυτό το ζήτημα της ανεργίας των νέων που μαστίζει όλη την Ευρώπη και για το φαινόμενο τέλος των φτωχών εργαζομένων που καθημερινά εξαπλώνεται. Θα ήθελα κλείνοντας να ευχηθώ ολόψυχα λόγω και των ισχυρών δεσμών που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μας κάθε επιτυχία και στην Κυπριακή Προεδρία αλλά και σε εσάς προσωπικά για την ιστορία σας που τη γνωρίζουμε όλοι. On va encore prendre deux. Δύο ακόμη ομιλητές να ακούσουμε. Κρίστενσεν και μετά Μόραν Σαρτιέ. Κρίστενσεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και την ε, κυρία Υπουργό για την παρουσίαση που μας έκανα. Ήσασταν πιστεύω ξεκάθαροι σε ό,τι αφορά την οδηγία για την ε, απόσπαση εργαζομένων Αλλά νομίζω ότι για τον κανονισμό Μόντι 2 έχω κάποιες αντιρρήσεις. Δίκαιο έχετε για την κίτρινη κάρτα από τα κράτη-μέλη, αλλά θα ήθελα να ακούσω πιο πολύ την δική σας άποψη για αυτόν τον κανονισμό. Σύντομο ήσασταν και πολύ ακριβής, η κυρία Μωράν Σαχτιέ. Ευχαριστώ πολύ, ε, κύριε Υπουργέ. Θα σας θέσω τρία ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ε, για το οποίο τοποθετηθήκαμε την περασμένη εβδομάδα εμείς ως Επιτροπή. Η ψηφοφορία της Επιτροπής μας ε, δείχνει ότι επιθυμούμε σε αντίθεση με το Συμβούλιο, 25% των ε, ταμείων συνοχής ε, να ε, είναι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ότι η ρήτερα μακροοικονομική επιλεξιμότητα να μην ισχύει για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να αποφύγουμε την ε, διπλή ε, τιμωρία των ε, μισθωτών και 20% του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου να αφιερωθεί στην καταπολέμηση της φτώχειας. Ποια είναι η δική σας άποψη για αυτά τα τρία σημεία τα οποία μας απασχολούν όλος ιδιαίτερος. Δεύτερο ερώτημα που θα ήθελα να σας θέσω αφορά τη νέα οδηγία για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία η οδηγία του 2004 συμπεριλάμβανε με καταχρηστικό τρόπο για να το πω έτσι, όλο τον ιατρικό εξοπλισμό και τις MRI, τις μαγνητικές τομογραφίες, ε, ποια είναι η άποψή σας, μήπως θα έπρεπε να ε, αναθεωρήσουμε το κείμενο ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν ε, στη διάθεσή τους αυτές τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, αφήνοντας βέβαια τις απαραίτητες διατάξεις για την υγεία των πολιτών. Ποια είναι η άποψή σας και πώς θα κινηθείτε επ' αυτού. Όσον αφορά τώρα την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, την αναφέρατε, μυρίσατε για την ίση αμοιβή. Εγώ θα ήθελα μία ακόμη φορά να σας ρωτήσω για την ισότητα στις καριέρες. Ε, ε, τι έχετε σκοπό να κάνετε. Είναι πολύ δυσκολότερες για τις ε, γυναίκες από ό,τι για τους άντρες και όπως επίσης και για την κοινοβότηση. Ευχαριστώ πολύ θα ήθελα να συμπληρώσω αυτό που είπε η κυρία Μωράν Σάτι, επειδή σας δώσω το λόγο, να σας πω ότι καταψήφισε την μακροοικονομική επιλεξιμότητα όχι μόνο για το Ευρωπαϊκό Κεντρικό Ταμείο η δική μας Επιτροπή, η κυρία Μωράν Σάτι ήταν η συγγήτρια, αλλά και για το γενικό κανονισμό. Δεν θέλουμε καθόλου αυτού του είδους την επιλεξιμότητα. Ε, την απόφαση λάβαμε ε, ε στην έκθεση του ε, συναδέλφου συναδέλφου μας. Νομίζω ότι είναι μια πιο οριζόντια, ένα πιο οριζόντιο ζήτημα ε, αυτό. Έχω να σας δώσω το λόγο και μετά να δώσω το λόγο σε άλλους πέντε ομιλητές. Ευχαριστώ. Ξεκινήσω την απάντηση μου από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, γιατί ήταν παράληψη μου στις προηγούμενες τοποθετήσεις υπήρχε ερώτημα και δεν το είχα απαντήσει. Λέγοντας ότι και στο θέμα το οποίο, που αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ο στόχος μας έχοντας υπόψη τη δουλειά που έχει γίνει επί Δανική προεδρία, που όπως έχω ήδη αναφέρει είναι, ήταν πάρα πολύ καλή και αξιόλογη και μα βοηθά να προχωρήσουμε παραπέρα είναι να ολοκληρώσουμε και να δώσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο που θα απαντά στον κεντρικό στόχο που έχει η οδηγία που είναι η προστασία και η ασφάλεια των εργαζομένων ε, από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ταυτόχρονα σε αυτή τη διαδικασία δεν μπορεί παρά να λάβουμε υπόψη και αυτό στο οποίο η κυρία Μωρίν έχει ε, αναφερθεί, δηλαδή ε, την, ανάγκη για χρήση της, ε, το, της μαγνητικής τομογραφίας στον τομέα της υγείας. Εμείς θεωρούμε ότι λαμβάνοντα υπόψη και τι ε, απόψει των ειδικών και εκείνων που έχουν την τεχνογνωσία και εγώ δεν είμαι ειδικό και δεν έχω την εξειδικευμένη τεχνογνωσία αλλά εν πάση περιπτώσει εκείνο το οποίο πρέπει να βρούμε είναι την ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας και της υγείας ε, των εργαζομένων και της ανάγκης ε, για χρήση αυτής της τεχνολογίας Μέσα σε ένα σωστό πλαίσιο. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα τα άλλα ερωτήματα να, για τα θέματα που έχουν εγερθεί ε, για το πρόγραμμα για την καινοτομία και την ε, κοινωνική αλλαγή και τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει από πλευράς του Ευρωκοινοβουλίου, τις παρατηρήσεις του Ευρωκοινοβουλίου. Ε, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια διαδικασία που μόλις τώρα έχει ολοκληρωθεί από την ε, δική σας ε, την πλευρά. Οι διαπραγματεύσεις τώρα, έχουν, τώρα μόλις ξεκινούν, επομένως δεν έχουμε εντολή ακόμα από το Συμβούλιο για το πώς θα κινηθούμε. Θα αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και μετά από τις θερινές διακοπές θα τις εντείνουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Στο σημείο αυτό εγώ θα ήθελα ιδιαίτερα να υπογραμμίσω την ανάγκη ε, αυτός ο κανονισμός ε, να γίνει με τέτοιο τρόπο έτσι που να εκπληρώνει το στόχο του και ο κεντρικός του στόχος πρέπει να είναι προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης, της απασχόλησης, της ε, κοινωνικής συνοχής και της ε, καινοτομίας. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι το καθοδηγητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο ε, πρέπει να, να κινηθούμε. Ε, σε ό,τι αφορά το ερώτημα που έχει τεθεί για τους ε, εργαζόμενους ε, σε παραμεθόριες περιοχές, θα επαναλάβω για ακόμα μια φορά την βασική αρχή κάτω από την οποία εμείς βλέπουμε να λειτουργεί το θέμα της κινητικότητας των εργαζομένων, που είναι η αρχή της ισότητας. Και προερχόμενοι από μια χώρα που έχουμε μεγάλο αριθμό ε, εργαζομένων από άλλες χώρες μέλη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχοντας τις δικές μας εμπειρίες θα ήθελα ιδιαίτερα να υπογραμμίσω την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και σε διμερές επίπεδο γύρω από αυτά τα, τα ζητήματα. Χρειαζόμαστε διαφάνεια, χρειαζόμαστε συνεργασία και αποτελεσματικούς εφαρμοστικούς μηχανισμούς για να μπορέσουμε να διασφαλίζουμε ε, τα, τα βασικά ζητούμενα γύρω από το πλαίσιο ε, της ε, διακίνησης των εργαζομένων. Κατανοώ, αντιλαμβάνομαι και πλήρως αποδέχομαι την έγνοια που όλοι έχουμε ειδικότερα οι ευρωβουλευτές που συμμετέχουν στην Επιτροπή Απασχόλησης ε, του Κοινοβουλίου για άμεσες λύσεις. Λύσεις οι οποίες θα απαντούν στα καυτά προβλήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα ως ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η Κυπριακή Προεδρία έχει αποφασίσει να εστιάσει την προσοχή της στα θέματα της ανεργίας ανάμεσα στους ε, νέους, πραγματοποιώντας και ειδικό συνέδριο προς ε, αυτή την ε, κατεύθυνση. Η δική μας η προσπάθεια είναι, αξιοποιώντας εκείνες τις πολιτικές και εκείνα τα εργαλεία τα οποία έχουμε, και ειδικότερα θα ήθελα να αναφερθώ στο πακέτο για την απασχόληση και το γεγονός ότι μέσα από το πακέτο για την απασχόληση δίνεται έμφαση σε τομείς της οικονομίας όπως η πράσινη ε, οικονομία, οι θέσεις εργασίας στον ε, τομέα της ε, υγείας, οι θέσεις εργασίας στην τεχνολογία της πληροφορικής δίνοντας έφαση λοιπόν στις προοπτικές αυτών των τομέων και πώς οι προοπτικές αυτών των τομέων διασυνδέονται με πολιτικές που θα οδηγούν σε θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχουν λύσεις οι οποίες μπορούν να δοθούν μόνο από το Συμβούλιο, όπως δεν υπάρχουν και λύσεις οι οποίες μπορούν να δοθούν μόνο από την Επιτροπή. Εκείνο το οποίο νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να εισάξουμε στην προσπάθεια για ανάπτυξη και ολιστικές πολιτικές οι οποίες να λαμβάνουν υπόψη από τη μια και είναι οι τομείς της οικονομίας που αυτή τη στιγμή παρουσιάζουν καλύτερες προοπτικές να διασυνδέσουμε αυτούς τους τομείς με τις, με τις εκπαιδευτικές πολιτικές αλλά και τις πολιτικές ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού για να, για οδηγηθούμε σε αυτό που είναι το κεντρικό ζητούμενο θέσεις εργασίας. Άρα εστιάζοντας σε αυτή την προτεραιότητα για την νεανική απασχόληση εμείς ταυτόχρονα θα δούμε όλες εκείνες τις παραμέτρους που επηρεάζουν την νεανική απασχόληση και με τον ίδιο φακό ε, θα δούμε και τις ε, παραμέτρους που αφορούν τα θέματα της ανασφάλισης της εργασίας. Είναι σημαντικό το ότι μέσα στο πακέτο για την απασχόληση υποδεικνύεται ή αν θέλετε υπογραμμίζεται το θέμα της αδήλωτης και παράνομης ε, εργασίας και ε, ακριβώς είναι και στα χέρια των κρατών μελών αλλά και μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών να προωθήσουμε εκείνες τις πολιτικές ε, που ε, θα καταπολεμήσουν το φαινόμενο της ανασφάλισης της εργασίας. Σε ό,τι αφορά την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και να μου επιτρέψετε να συνδέσω την απάντησή μου σε αυτό το ερώτημα με τα ερωτήματα για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο η διαπραγμάτευση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου ε, θα γίνει σε ένα άλλο πλαίσιο. Είναι κομμάτι της διαπραγμάτευσης για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Εκείνο το οποίο θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι από την πλευρά της Κυπριακής Προεδρίας ε, θεωρούμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ω ένα σημαντικότατο εργαλείο στην διαδικασία για πρόθεση της ανάπτυξης που δημιουργά θέσεις εργασίας και στη διαδικασία της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα φροντίσουμε έτσι που το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να έχει εκείνο το βάρος μέσα στον προϋπολογισμό της Ένωσης για τα επόμενα χρόνια που θα το επιτρέψουν να παίζει αποτελεσματικά αυτό το ρόλο και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι θα διαβιβάσω τα ζητήματα τα οποία μας έχετε θέσει τόσο εσείς κυρία ε, Πρόεδρο όσο και η κυρία Μωρήρη στην ομάδα της ε, Κύπρου που θα διαπραγματευτεί το ε, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Για τον κανονισμό Μόντι 2 ήταν ένα άλλο ερώτημα που μου έχει τεθεί ως ε, πρόεδρος του Συμβουλίου δεν μπορεί παρά να περιμένουμε την ε, θέση της, ε, της Επιτροπής. Εκείνο που θα ήθελα να σας πω σε προσωπικό επίπεδο ως Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου είναι ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτή τη διαδικασία να φροντίσουμε έτσι που βασικά θεμελιώδη δικαιώματα όπως το δικαίωμα της συλλογικής δράσης λαμβάνοντα υπόψη ότι οι εθνικέ πρακτικές και οι εθνικέ νομοθεσίε αυτό το θέμα το χειρίζονται με διαφορετικό τρόπο να ληφθεί υπόψη σε όλη αυτή την, ε, ε, διαδικασία. Θα περιμένουμε την Επιτροπή και νομίζω ότι έχοντας όλοι εμπειρίες και έχοντας υπόψη και τις εθνικές ιδιαιτερότητες ε, θα βρούμε εκείνες τις λύσεις που θα διασφαλίζουν ότι προχωρούμε μπροστά. Για τα θέματα της ισότητας ε, στην, ε, ε, καριέρα. σαφέστατα έχει τεράστια σημασία τόσο η διασφάλιση της ίσης αμοιβή, αλλά και οι πολιτικές που βοηθούν τις ε, γυναίκες να μπορούν να είναι στην αγορά εργασία με προοπτικές και με φιλοδοξίες, με τη θετική έννοια και με επιδιώξεις. Θα έλεγα ότι αυτά τα ζητήματα χρειάζονται ένα πλέγμα από πολιτικές. Δεν είναι ζητήματα τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσα από νομοθετικές πρωτοβουλίες ή μόνο μέσα από τις πολιτικές απασχόλησει. Είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες οι οποίοι επιδρούν. Το πρωί είχαμε την ευκαιρία μαζί με τον συνάδελφο Υπουργό Δικαιοσύνη και Δημόσια Τάξη, που είναι ο υπεύθυνο Υπουργό για θέματα ισότητα στην Κύπρο, να παρευρεθούμε στην Επιτροπή Ισότητα του Ευρωκοινοβουλίου και εκεί έχουμε υπογραμμίσει ότι τα θέματα της ισότητας είναι πολύ σημαντικά για την Κυπριακή Προεδρία. Εξού και πέραν από το θέμα της ίσης αμοιβή έχουμε θέσει ως προτεραιότητα μας και τα θέματα της ε, βίας ενάντια στις ε, γυναίκες. Εκείνο που θα ήθελα να πω για το θέμα που έχετε θίξει είναι το εξή. Χρειάζεται μέσα από τις πολιτικές απασχόλησεις να συνεχίσουμε να δίνουμε έμφαση στην απασχόληση των γυναικών. Και όταν λέω στην απασχόληση των ε, γυναικών, θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό και την ποιότητα της απασχόλησης των γυναικών. Ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα σημαντικό μέσα από τις πολιτικές που εφαρμόζουμε και σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει να παίξει τον δικό του ρόλο στα θέματα της ισορροπίας μεταξύ οικογένειας και εργασίας. Ε, ταυτόχρονα όμως ε, υπάρχουν και πολιτικές τις οποίες μπορούμε να αξιοποιήσουμε όπως την πρωτοβουλία για τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ειδικότερα στα θέματα της συμμετοχής τους στα συμβούλια των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ράπτη και μετά η κυρία Βνικεβιτσιούτη. Κυρία Ράπτη πρώτα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλωσορίζω την Υπουργό. Μου αρέσει που είναι εδώ Υπουργό Εργασίας και μάλιστα γυναίκα. Ε, αυτό μας κάνει να ελπίζουμε περισσότερα. Είπατε κυρία Υπουργέ ότι οι λύσεις δεν θα έρθουν μόνον από το Συμβούλιο ή μόνον από την Επιτροπή. Να προσθέσω ότι οι καλύτερες λύσεις έρχονται όταν συμμετέχει το Κοινοβούλιο. Και να περάσω σε δύο θέματα το ένα είναι και πάλι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ε, δεν μπορώ να αποφύγω τον πειρασμό να επανέλθω σε αυτό το θέμα δεδομένου ότι είμαι σκιώδης εισηγήτρια από την πλευρά των σοσιαλιστών και δημοκρατών για το θέμα. Ε, θα βάλω το εξής πολύ συγκεκριμένο ερώτημα ε, δεδομένου ότι τα υπόλοιπα καλύφθηκαν από τους καλούς συναδέλφους που αφορά την επίπτωση της χρήσης των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στους εργαζομένους. Εδώ έχουμε δύο πράγματα. Τις μακροχρόνιες επιπτώσεις και τις βραχυχρόνιες επιπτώσεις. Ωστόσο δεν έχουμε επιστημονικές μελέτες που να τεκμηριώνουν ότι η επαναλαμβανόμενη βραχυχρόνια έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία επιφέρει βλάβες ή όχι. Υπό αυτήν την έννοια εμείς έχουμε στο μυαλό μας ως σοσιαλιστές, ως ομάδα σοσιαλιστών και δημοκρατών ε, το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεχής επιστημονική έρευνα σε σχέση με αυτό το ζήτημα και ρωτώ εάν είναι στις προθέσεις σας, εάν είναι στις σκέψεις σας να βάλετε και αυτή τη διάσταση στην πρότασή σας. Το δεύτερο ζήτημα είναι η υπεργολαβία. Είναι ένα θέμα για το οποίο δεν υπάρχει νομοθεσία όπως ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα. Και το ερώτημα είναι είστε διατεθειμένοι ως Κυπριακή Προεδρία πια να το προχωρήσετε αυτό το θέμα. Θα εξετάζατε το ενδεχόμενο να ζητήσετε από την Επιτροπή να διερευνήσει τις δυνατότητες για έναν ευρωπαϊκό νόμο σε σχέση με τις αλυσιδωτές ευθύνες στο θέμα της υπεργολαβίας. Ταλαιπωρούνται πάρα πολλοί εργαζόμενοι σε ολόκληρη την Ευρώπη από αυτή την υπόθεση. Και κλείνω, κυρία Πρόεδρε, για να είμαι σύντομη, ε, δύο θέματα το πρώτο είναι ότι προσωπικά επιτρέψτε μου να τρέφω πολλές ελπίδες ότι η κυπριακή προεδρία θα είναι αποτελεσματική. το δεύτερο είναι ότι καλύφθηκα ως γενική τοποθέτηση και γι' αυτό δεν την επαναλαμβάνω από την τοποθέτηση που έκανε ο καλός έλληνας συνάδελφός μου που ανήκει ε, στο ΕΠΠ ο κύριος πουπάκης και αυτό νομίζω ότι σας δίνει μια εικόνα για την προσπάθεια που κάνουμε και εδώ στο κοινοβούλιο για τα θέματα της απασχόλησης και της αντιμετώπισης της ανεργίας και της φτώχειας αλλά και την προσπάθεια που προσπαθούμε να κάνουμε ως ελλάδα που πλήττεται βαρύτατα αυτό τον καιρό. σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία και μετά η κυρία Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ. Αναλαμβάνετε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια δύσκολη χρονική στιγμή, όταν όλη η Ευρώπη βρίσκεται βαθιά σε μια οικονομική κρίση, κάτι που έχει επηρεάσει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων και στα καθήκοντά σας, βεβαίως, έχετε και τις επραγματεύσεις για το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο έως το 2020. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, να έχετε ένα συνεχή διάλογο με μας ε, στο Ευρωκοινοβούλιο για αυτά τα θέματα. Κάποιες τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αν προκειμένου είναι και αρκετά δυσνόητες για μας, ειδικά τη συμπερίληψη της γεωργίας στο Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί η Κυπριακή Προεδρία θα εστιάσει στα θέματα της φτώχειας και του ε, κοινωνικού αποκλεισμού και μπορώ να το επικροτήσω αυτό ιδιαίτερος, διότι πολλοί άνθρωποι ακόμη βιώνουν την φτώχεια και το κοινωνικό αποκλεισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πιο αποτελεσματικό τρόπο, πιστεύω, για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων είναι η απασχόληση, η δημιουργία θέσεων εργασία. Είπατε ότι και εσείς και η, Ισπαν... και η Κυπριακή Προεδρία θα εστιάσει στις ποιοτικές σας εργασίες, όχι απλά στη δημιουργία της εργασία, αλλά στην ποιότητα. Θέλω λοιπόν να σα ρωτήσω τι συγκεκριμένα μέτρα έχετε στο μυαλό σα να προωθήσετε κατά τη διάρκεια τη Προεδρία σα για ποιοτική ε, εργασία και πώ θα το συνδέετε με το flexicurity, την ευελιξία και την ασφάλεια στην εργασία. Πώς δηλαδή μπορούμε να ισορροπήσουμε μεταξύ των δύο. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να επισημάνω. Θα γνωρίζετε βεβαίως ότι υπάρχουν και άνθρωποι που εργάζονται, που είναι στην εργασία, αλλά παρόλα αυτά βρίσκονται στη φτώχεια, διότι ε, πολλές φορές οι αμοιβέ πέφτουν πάρα πολύ χαμηλά. Ε, είναι θέματα τα οποία ε, σκοπεύετε να προωθήσετε με κάποιες προτάσεις. Και επίσης για τις συντάξεις. Το στεξιωτικό θέλω να θέσω ένα ζήτημα. Ξέρετε, υπάρχουν συγκεκριμένες ε, συστάσεις ε, για την διασφάλιση επαρκών και αξιοπρεπών συντάξεων. Ε, αλλά, να ρωτήσω το εξή. Πολλά κράτη-μέλη έχουν αυξήσει το όριο συνταξιοδότησης, το ηλικιακό όριο, ε, αλλά ταυτόχρονα δεν βλέπω αντίστοιχα μέτρα που να προωθούν την απασχολησιμότητα ανθρώπων σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ρωτώ, αν είναι κάτι που σας απασχολεί και εσάς και τι θα κάνετε σχετικά με την απασχολησιμότητα ε, ανθρώπων μεγαλύτερων ηλικιών. Και κάτι ακόμη. Να σας ευχαριστήσω θερμά για τις έως τώρα πολύ καλές απαντήσεις που μας έχετε δώσει. Μία ακόμη συμπληρωματική ερώτηση, κυρία Τσούμπερ. Ε, πρώτα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Υπουργό για την παρουσία της στην Επιτροπή μας. Και θέλω να πω ότι παρατηρώ με ιδιαίτερη ικανοποίηση την παρουσίαση που κάνατε καθώς προσπαθήσατε με οριζόντιο τρόπο να μιλήσετε για την κοινωνική προστασία και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. πολύ συχνά σε αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε για τα δημοσιονομικά ξεχνούμε αυτά ακριβώς τα θέματα που εσείς θέσατε. Εμείς θέλουμε ειδικά να εστιάσουμε την προσοχή στις θέσεις εργασίας, αλλά κάνουμε πρώτα απ' όλα ένα σχόλιο. Μιλούμε για τη δημιουργία θέσεων εργασίας ως ζωτική σημασία για την ίδια την οικονομία, αλλά και για την κοινωνική πρόοδο και για την βελτίωση του βιωτικού επίπεδου όλων. Ωραία. Μιλούμε λοιπόν εργασία. Δεν μιλούμε όμως ταυτόχρονα και για την α, κατάργηση και την απώλεια θέσεων εργασίας. Έχει νόημα να μιλούμε για τη δημιουργία θέσεων εργασία όταν παραγνωρίζουμε το πρόβλημα της απώλειας, της καταστροφής. Μιλάμε για πολλές φορέ για μαζική καθημερινή απώλεια θέσεων εργασία. Τόσο ένα παράδειγμα από τη χώρα μου, όπου εδώ και ένα χρόνο Χάραμε καθημερινά 558 θέσει εργασία. Καθημερινά το τελευταίο έτος. Μιλάμε για έναν αγώνα ταχύτητας απώλεια θέσεων εργασία. Μιλούμε λοιπόν συνεχώς για δημιουργία νέων θέσεων. Ναι, πρέπει ταυτόχρονα να διαφυλάξουμε και τις υπάρχουσες θέσει εργασία. Αυτό πρώτα απ' όλα θέλω να θέσω. Θα πρέπει λοιπόν να επισημάνουμε τις την πολύ αρνητική, με τον αρνητικό αντίκτυπο των πολιτικών ε, που, στο οποίο καταθέτουν πολλές κυβερνήσεις, την απόλυση δημοσίων υπαλλήλων. Υπάρχει βεβαίως στον ειδικό τομέα και το σοβαρό πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας της επιχειρήσης, οπότε αναγκάζονται πολλές επιχειρήσεις να βάλουν κέτο ή να απολύσουν μαζικά προσωπικό. Και θα ήθελα να πω ότι όχι μόνο πρέπει να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις σε όλα τα επίπεδα, ιδίω οι μικρομεσαίες, αλλά θα μιλούσα και για ανάγκη αύξησης ε, των μισθών για να μπορεί να στηριχθεί ο κοινωνικός ιστός. Έπειτα, οι απολύσεις και κατάργηση τη εργασίας, όλα αυτά που οδηγούν στην αλλίωση ε, των εργασιακών δικαιωμάτων και του εργατικού δικαίου, οδηγώντας σε όλο και πιο φθηνή απασχόληση. Λοιπόν, δεν πρέπει να περιορίζουμε τη συζήτηση στην δημιουργία νέων θέσεων εργασία. Αν δεν δούμε ποια είναι τα αίτια που οδηγούν στην απώλεια τόσων θέσεων εργασία, πιστεύω ότι αλλιώ περιοριζόμαστε σε μία ατέρμονα συζήτηση που είναι ελάχιστα παραγωγική. Έπειτα, η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ε, μέσω προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα τα EURES και τέτοια ε, αντίστοιχα προγράμματα πολύ σημαντικά για την προώθηση απασχόληση, ότι είναι ζωτική σημασία θα έλεγα μάλιστα ότι θα πρέπει να ενισχυθεί όχι μόνο ο συνολικός προπολογισμό του, του Κοινωνικού Ταμείου, αλλά και του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού εν γέννη, για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε όλες τις χώρες της Ένωσης, ιδίως τις πλέον αδύναμες ε, χώρες αυτή τη στιγμή οικονομικά, αυτές που επηρεάστηκαν περισσότερο αρνητικά από την εφαρμογή της, της ε, ολοκλήρωσης αγοράς. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, πρέπει να αντιστρέψουμε αυτή τη διαδικασία που αφορά την απασχόληση ένα φαινόμενο όλο και πιο συχνό. Χάνονται, χάνονται συνέχεια θέσεις εργασίας, κυρίως για άτομα με μεγάλη προπηρεσία, προπηρεσία 30 και άνω ετών, Διακόπτη Πρόεδρος, ζητώντας ε, να μην μακρηγορεί ο Μιλήτρια. Ναι, ναι, βεβαίως. Συνεχίζει ο Μιλήτρια. Αντικατάσταση λοιπόν της εργασίας, μάλλον απολύονται εργαζόμενοι με μακρά ε, προϋπηρεσία και αντικαθίστανται με νέους εργαζόμενους μεν, αλλά με πολύ πιο χαμηλές απολαβές, με πολύ λιγότερα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα και λιγότερη γενικότερη ασφάλεια στην εργασία. Η απασχόληση για τους νέους δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτό το δρόμο δεν είναι αυτό ένα παράδειγμα προ μίμηση, δεν ήταν αυτό που είχαμε ποτέ στο μυαλό μα όταν μιλούσαμε για κοινωνική πρόοδο για του εργαζόμενου και για την ανθρωπότητα εν γέννη. Μας ανησυχεί λοιπόν ιδιαίτερα το γεγονό ότι σε πολλέ χώρες Κυρία Τσούμπερ, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γιαζουοβιέτσκα αλλά σας ζητώ πρώτα να είστε πάρα πολύ σύντομοι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλήσουν και οι υπόλοιποι και να έχει και τη δυνατότητα η υπουργό να απαντήσει, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε με αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Κυρία Γιαζιοβιέτσκα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω τις ευχαριστίες μου ε, στην Υπουργό για τις προτεραιότητες ε, της Κυπριακής ε, Προεδρίας, τις οποίες μας παρουσίασε. Μιλήσατε για την υποστήριξη των αποσπασμένων εργαζομένων. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια ζητήματα είναι ευαίσθητα ή αντιφατικά στο Συμβούλιο για αυτό το θέμα, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Εμείς ψηφίσαμε τον κανονισμό την περασμένη εβδομάδα. Πολλές φορές ακούμε αρνητικές απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το Ταμείο, όπως επίσης και για την αποτελεσματικότητα ε, των θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται και τη σταθερότητα αυτών. Εμείς ψηφίσαμε 25% το προορισμού να πηγαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Σε κάποιες χώρες όμως ε, υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης ε, τέτοιων δραστηριοτήτων. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε αυτό το 25% το ελάχιστο. Ποια είναι η άποψη των περισσότερων κρατών μελών για το θέμα αυτό. Θα χρησιμοποιηθεί επαρκώς ε, και σωστά το Ταμείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Νταρντένα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος γιατί υπήρξαν ήδη πολλές ερωτήσεις και τα θέματα τα οποία ήθελα να θέσω κι εγώ κάπως καλύφθηκαν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Υπουργό για την παρουσίασή της, την παρουσία, την της, την παρουσίασή της και τις απαντήσεις της και όπως ε, υπόθηκε και στην Ολομέλεια του Στραβούργου, όπως ε, οι βασικές προκλήσεις για το μέλλον θα είναι το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τα διαρθρωτικά ταμεία. Ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα διαρθρωτικά ταμεία να εξακολουθούν να καλύπτουν το σύνολο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιμένω στη σημασία ε, των ε, ταμείων αυτών, ειδικότερα στις περιφέρειες. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας γι' αυτό. Ξέρω ότι δεν ε, είναι αντικείμενο ομοφωνίας, αλλά θα ήθελα να ακούσω την άποψη της Προεδρίας. Υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και είναι σημαντικό να πρικοδοτηθεί με αρκετά καλό τρόπο ώστε να μπορέσει να βοηθήσει στην καταπολέμηση της ένα ακόμη κοινωνικό στοιχείο ε, αφορά το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω την άποψή σας για τη δυνατότητα ε, της αναδιάρθρωσης και της χρήσης της με ευρύτερο τρόπο από ότι... Τη ε, γίνεται ως τώρα. Υπάρχουν κάποια μέλη του Συμβουλίου που θέλουν να εξαφανιστεί. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω την άποψή σας για το θέμα τώρα των συντάξεων. Ξέρω και πάλι ότι κάποια μέλη του Συμβουλίου ε, συμφωνούν με την αύξηση της ταξιοδότησης που έχει να κάνει με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Νομίζω ότι είναι μία λανθασμένη άποψη. Ε, νομίζω ότι πρέπει να αυξήσουμε την ε, ε ενεργό ηλικία ε, έναρξης επαγγελματικού βίου για να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε το ποσοστό απασχόλησης σε διάφορες κατηγορίες, μεταξύ των νέων για παράδειγμα, να αυξηθεί η απασχόληση. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας και για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Υπουργέ, θα ήθελα να σας ζητήσω να απαντήσετε σύντομα στις ερωτήσεις αυτές. Νομίζω ότι ήταν ένας τρόπος να σφιγουμετρήσετε και την άποψη των μελών της Επιτροπής μας και να ξέρετε τα θέματα που θα πρέπει να διαπραγματευτούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανταποκρινόμενη στην παράκληση σας, θα προσπαθήσω να κάνω κάποια γενικά σχόλια και να πω ότι για ειδικά ερωτήματα που έχουν τεθεί είτε σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία είτε για άλλα ειδικά ερωτήματα θα επανέλθουμε με, ε, με γραπτές ε, απαντήσεις για να μπορέσουμε να κερδίσουμε κάποιο χρόνο. Ε, νομίζω ότι από τα ερωτήματα και από τη συζήτηση έχει αναδειχθεί πόσο οι πολιτικές οι οποίες ακολουθούμε έχουν το στοιχείο της αλληλοεπίδρασης και της αλληλοσυμπλήρωσης. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τις ε, πολιτικές απασχόλησης και τις πολιτικές για καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Είναι σημαντικό να στηρίξουμε την προσπάθεια για να έχουμε θέσεις εργασίας, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να στηρίξουμε την προσπάθεια για να έχουμε τους διαθέσιμους πόρους, για να δίνουμε ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας σε εκείνους τους πολίτες της Ένωσης που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ευελιξίας και της ασφάλειας. Εμεί θεωρούμε ότι η απάντηση είναι στην ισορροπία. Η δυνατότητα ειδικότερα μέσα από τον κοινωνικό διάλογο μέσα από τις εθνικές πρακτικές που έχει η κάθε χώρα σε ό,τι αφορά τον οργανωμένο διάλογο συντεχνιών και εργοδοτών να βρίσκει λύσεις τόσο στο επίπεδο των επιχειρήσεων όσο και στο επίπεδο κλάδων οικονομικής δραστηριότητας που να ανταποκρίνονται στις σημερινές δύσκολες συνθήκες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έρχεται σε αντιδιαστολή και να θέτει υπό αφισβήτηση τα δικαιώματα των εργαζομένων τα δικαιώματα των εργαζομένων όπως απορρέουν και από οδηγίες και νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω από το ίδιο πλαίσιο αντιμετωπίζουμε και το θέμα της υπεργολαβίας. Ανεξάρτητα από τη μορφή της εργασίας, τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σχέση εργοδότη-εργοδοτούμενου και τα οποία σε πολλές περιπτώσεις μέσα από οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελούν εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών διασφαλίζονται, πρέπει σαφέστατα οι χώρες να έχουμε τους μηχανισμούς για να μπορέσουμε να εφαρμόζουμε αυτά τα οποία είναι υποχρέωση και δέσμευσή μας έναντι ε, του κοινοτικού δικαίου. Σε ό,τι αφορά τα θέματα των συντάξεων, και ε, τα θέματα που αφορούν ε, την ε, επέκταση του εργασιακού βίου. Και εδώ θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά λέγοντας ότι σαφέστατα και από την πλευρά της Επιτροπής και από την πλευρά του Συμβουλίου έχουν υπάρξει αρκετές πρωτοβουλίες πρόσφατα. Το Συμβούλιο μας έχει υιοθετήσει συμπεράσματα γύρω από τα θέματα των συντάξεων. Ο κεντρικός στόχος πρέπει να είναι η βιωσιμότητα αλλά και η επάρκεια των συντάξεων. Και έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία πρέπει να σα πω για τα θέματα των συνταξιούχων γιατί η Κύπρο είναι μια από τι χώρε που έχει ψηλό επίπεδο φτώχεια ανάμεσα στου συνταξιούχου. Μειώνεται αλλά εξακολουθεί να είναι ψηλό. Και θα έλεγα ότι έχουμε μια ιδιαίτερη υποχρέωση σε αυτή την γενιά των Ευρωπαίων πελετών να του διασφαλίσουμε επάρκεια σύνταξη. Οι τρόποι που θα διασφαλίσουμε αυτά αυτές τις δύο βασικές αρχές είναι στα κράτη-μέλη, διότι είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών να βρουν εκείνες τις πολιτικές οι οποίες θα συνάδουν με τα δικά τους δημογραφικά και οικονομικά δεδομένα. Θέλω όμως ιδιαίτερα να υπογραμμίσω την ανάγκη να έχουμε πολιτικές, και αυτό συνδέεται με τις πολιτικές απασχόλησης και τις πολιτικές κατάρτισης, έτσι που οι εργαζόμενοι μέσα από συνεχή διαδικασία κατάρτισης και επανακατάρτισης να αποκτούν ευκαιρίες για παραμονή στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι, αυτό είναι και το σημαντικό ζήτημα όταν μιλούμε για την επάρκεια ε, των ε, συνταξιδοτικών ε, δικαιωμάτων και για την επέκταση του εργασιακού βίου που με τη σειρά του έχει τη δική του επίδραση και στα ζητήματα της βιωσιμότητας ε, των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ερωτήματα. Αντιλαμβάνομαι ότι ο, χώρος, ο χρόνος μας έχει ε, λήξει. Ε, εκείνο που θα ήθελα να, να σας πω ε, ολοκληρώνοντας είναι ότι για μένα και για τους συνεργάτες μου από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι επισημάνσεις σας, οι παρατηρήσεις σας, οι εισηγήσεις σας είναι πάρα πολύ σημαντική στη διαδικασία που θα έχουμε μπροστά μας και σαφέστατα θα μπορέσουμε να έχουμε το χρόνο στην Κύπρο να συζητήσουμε και συγκεκριμένα ζητήματα που δεν είχαμε το χρόνο να τα καλύψουμε τώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ θα βρεθούμε σε δύο μέρες ε, στη Λευκοσία, ε, στο ε, Συμβούλιο και ούτως ή άλλως θα έχουμε τη δυνατότητα να σας ξαναδούμε στο τέλος Αυγούστου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα μας είπατε. Καταλαβαίνω ότι έχετε πολλή δουλειά. Ε, θα προσπαθήσουμε να σας ε, βοηθήσουμε ως Επιτροπή, διότι ε, συμφωνούμε, αν συμφωνούμε με τους προσανατολισμούς του Συμβουλίου, που θεωρούμε ότι θα ισχύσει για τα περισσότερα θέματα. Καλή τύχη και καλή επιτυχία. Chers collègues, nous en venons, Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε τις εργασίες μας και πάμε στο σημείο 21. Παρακαλώ λίγη ησυχία. Όσοι θέλουν να αποχωρήσουν, να αποχωρήσουν, αλλά ήσυχα, ώστε η κυρία Κίνγκα Γκούντς η συντάκτρια γνωμοδότησή μας, γνωμοδότησής μας να μπορεί να πάρει το λόγο και να μας παρουσιάσει τις τροπολογίες στο σχέδιο γνωμοδότησής της για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να σας πω ότι το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη έρχεται ως επιστέγαμα τη στέγασμα συγγνώμη, των δύο προηγουμένων προγραμματών, το Europa Mundis και αυτό οφείλεται βεβαίως ε, στο υψηλό ύψος των κοντιλίων που δίνονται σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Έχουμε να κάνουμε με ένα σημαντικό τομέα. Ένα σημαντικό τομέα γιατί βοηθά στη δημιουργία θέσεων εργασία. Πρέπει λοιπόν να προσαρμοστεί αυτός ο, ο τομέας τις νέες συνθήκες της παγκοσμιοποίησης και ούτω καθεξής. Συνολικά υπευλήθησαν 38 τροπολογίες από 7 μέλη της Επιτροπής μας, σχεδόν από όλες τις πολιτικές ομάδες και εστιάζουν κυρίως σε αυτά δημιουργική τομή, στη δημιουργικότητα γενικότερα για την ε, περισσότερη συμμετοχή στην ε, ε, ανάπτυξη, διευκόλυνση στην πρόσβαση σε ευκαιρίες, επαγγελματική κατάρτιση από εμάς από το ΕΛΚΑ, κινητικότητα στον πολιτιστικό τομέα τους πράσινους, προσοχή ιδιαίτερα στις ιδιαιτερότητες του, του πολιτισμού άρση των γλωσσικών φραγμών και δημιουργία θέσεων εργασία με την εφαρμογή του προγράμματος που θα συνοδευτεί από έναν διάλογο όλων των ενδιαφερομένων μερών. Επίσης έχουμε και κάποιες τροπολογίες για τις δυνατότητες που μπορούν να δώσουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις για τους νέους επιχειρηματίες και τη δημιουργικότητα στο επιχειρήν γενικότερα για άτομα που προέρχονται από μειονεκτικό περιβάλλον. Έπειτα, ο ρόλος των περιφερειών που έχουν άνισες ε, συνθήκες, όμως θα πρέπει να ζητούν ευκαιρίες για να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση ε, σε πιθανούς πελάτες. Λοιπόν, αρχίσαμε να δουλεύουμε με τις ε, τροπολογίες ώστε να βρούμε κάποιους συμβιβασμούς Θα σας δώσουμε αυτούς τους συμβασμού μόλις οριστικοποιηθούν. Λοιπόν, θα έχουμε μία συνάντηση των σκιωδών αρχές Σεπτέμβρη, καθώς αυτή είναι και η τελευταία εβδομάδα των εργασιών ουσιαστικά και όλες ψηφοφορίες έχουμε. 19 Σεπτεμβρίου η ψηφοφορία προβλέπεται για την Επιτροπή. Αυτά προς το παρόν. like any, any Παρακαλώ, αν υπάρχουν βεβαίω σχόλια, είμαι στη διάθεσή σας. Αν όχι, θα σας αποστείλουμε τις συμβαστικές τροπολογίες και θα τις συζητήσουμε το φθινόπωρο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς να πάρει το λόγο? Κύριε Μπέκερ. Ευχαριστώ πολύ. Die Qualität der Zusammenarbeit äh, äh, als Schattenberichterstatter mit der Berichterstatterin und dem Kreis der anderen äh, und insbesondere hervorheben, dass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 Οπότε, Όλο το καλοκαίρι έχετε στη διάθεσή σα για να μα στείλετε συμβιβαστικέ τροπολογίε. 17 Σεπτεμβρίου θα τι εξετάσουμε για να τι ψηφίσουμε την επομένη. Κάτι το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα και στην Επιτροπή Πολιτισμού να τις λάβει υπόψη, να λάβει υπόψη την γνωμοδότησή μας ε, κατά την ε, σύνταξη της ε, εκθεσής της. Πάμε στο 19 τώρα της ημερήσιας διάταξης και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Μπλίνκεβιτσούτε για την εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησή της ε, στο, Erasmus, ε, στο, πρόγραμμα στο Erasmus για όλους, στο πρόγραμμα της Ένωσης για την Παιδεία, την επαγγελματική κατάρτιση, την νεολαία και τον αθλητισμό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Στι επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές 2014 με 2020 προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουμε ένα ενιαίο πρόγραμμα που θα λέγεται έρασμο για όλους Το συνολικό ποσό που προτείνεται είναι 19 δισεκατομμύρια ευρώ και αν εγκριθεί σημαίνει ότι αυτό το ποσό θα είναι 17% ε, υψηλότερο σε σχέση με αυτό ε, που έχουμε αυτή τη στιγμή, κάτι το οποίο νομίζω ότι μπορεί να μας ικανοποιεί και έχει ε, αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε ως Επιτροπή είναι να προτείνουμε κάποιες τροπολογίες σε σχέση με την απασχόληση. Άλλα στοιχεία θα καλυφθούν από τις άλλες τέσσερις κοινοβουλευτικές ε, επιτροπές. Εμείς προτείνουμε να καλυφθούν τα εξής. Το, το όνομα του προγράμματος υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις η αρμόδια εισηγήτρια, η κυρία Ντόρις Πακ, συμφωνεί με το προτινόμενο όνομα. Δεν νομίζω ότι εμείς θα έπρεπε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Καλύτερα θα ήταν να επικεντρωθούμε στο περιεχόμενο και όχι στο όνομα. Πρέπει να επικεντρωθούμε στην σαφή δομή του και στην, ε, στον επιμερισμό της χρηματοδότησης, που επίσης πρέπει να είναι σαφής. Γι' αυτό το λόγο δεν προτείνω ένα ε, όνομα ως εναλλακτική λύση και σε σχέση τώρα τα επιμέρους προγράμματα, ναι, βεβαίως να προτείνουμε κάποια ονόματα και εμείς και μπορεί η Επιτροπή ε, Πολιτισμού να λάβει υπόψη στη συνέχεια τις προτάσεις μας. Κάποιες πτυχές έχουν να κάνουν ε, με την ενίσχυση των σχέσεων ε, της απασχόλησης και της εκπαίδευσης, ε, όπως επίσης και της απασχόλησης με τη μείωση της φτώχειας. Δεν έχουμε λοιπόν μόνο σκοπό να εφαρμόσουμε τους στόχους της Ευρώπης 2020, Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αλλάξει και η διάρθρωση του κανονισμού, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τώρα κάτι ένα τμήμα για τις δραστηριότητες για την νεολαία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Και εγώ προτείνω τις δραστηριότητες για τους νέους να τις ξεχωρίσουμε. Για την κατάρτιση και την εκπαίδευση θα μπορούσαμε να επικεντρωθούμε σε μερικούς επιμέρους τομείς, που είναι σημαντική για την Επιτροπή Απασχόλησης, να μιλήσουμε για παράδειγμα για τη διαβίου εκμάθηση, ε, για την, εκμάθηση των, ε, για την ε, εκπαίδευση των ενηλίκων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στην υποστήριξη της ανώτερης εκπαίδευσης Κάποιες οργανώσεις ε, όμως ε, ε, εκπαιδευτικές λένε ότι αυτό δεν είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλούν για την καταπολέμηση της ανεργίας στα έγγραφά τους και γι' αυτό θα έπρεπε να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν να προσελκύσουμε και νέους και ηλικιωμένους σε εξυγχρονισμένη διαβίου εκμάθηση και να προωθήσουμε μια κουλτούρα διαβίου εκμάθησης. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στους επιμέρους τομείς της εκπαίδευσης και να αναφερθούμε στους συγκεκριμένους στόχους. Όσον αφορά τώρα την κινητικότητα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών ε, σε σχέση, για παράδειγμα, με ε, την ε, εκμάθηση, την εκπαίδευση των νέων, Για ποιο λόγο η ανταλλαγή φοιτητών και διδασκόντων αφορούν μόνο την ανώτερη εκπαίδευση, μας ερωτούν αλλά δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα στους ε, άλλους τρόπους ε, εκπαίδευσης, όπως η διαβίου εκμάθηση και η εκμάθηση, η, η εκπαίδευση των ενηλίκων. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα έπρεπε να υπάρξουν τροπολογίες για το άνοιγμα αυτής της δυνατότητας σε όλους τους τομείς ε, κατάρτισης. Όσον αφορά τώρα τον προϋπολογισμό, υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να συζητήσουμε. Βάσει της πρότασης του Ευρωπαϊ... της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο καλούνται να αποφασίσουν μόνο για το 56% του συνολικού προϋπολογισμού. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δυσκολεύομαι να το καταλάβω. Για ποιο λόγο ο νομοθέτης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν μπορεί να αποφασίσει για παραπάνω από το ίμιση του προϋπολογισμού. Δηλαδή το υπόλοιπο ίμιση του, του προπολογισμού, τι θα κάνει, θα το κατανείμει κατά το δοκούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, δεν μπορεί να πει τίποτα. Άρα εγώ προτείνω να φτάσουμε μέχρι το 81% αντί για 56%, ίσως να υπάρξουν και άλλες εναλλακτικέ προτάσεις. Αλλά η δική μου πρόταση θα ήταν περισσότερο να, να διαθέσουμε στη διαβίου εκμάθηση και ε, στην εκπαίδευση και κατάρτιση των ε, ενηλίκων. Αν δούμε την ε, γυράσκουσα δημογραφική τάση, είναι και πιο λογικό να γίνει κάτι τέτοιο. Όχι μόνο 2% του προπολογισμού να πηγαίνει ε, σε αυτή την κατηγορία. Επόμενο ζήτημα έχει να κάνει με τις, τους εθνικούς φορείς που θα διαχειριστούν το πρόγραμμα αυτό. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν πόσους ε, συντονιστικούς φορείς και εθνικές υπηρεσίες θα ήθελαν να έχουν σε εθνικό επίπεδο. Ε, κάποιο κράτο μέλος μπορεί να, να, ε, μπορεί να αρκεστεί σε έναν, κάποια κράτη-μέλη μπορεί να χρειάζονται περισσότερους φορείς. Αυτό θα έπρεπε να είναι στη διακριτική ευχαίρεια του κράτους μέλους. Σε σχέση τώρα με το πρόγραμμα Ζωμονέ, μόνο δύο Ινστιτούτα αναφέρονται σε σχέση με τα προηγούμενα έξι. Μπορώ να συμφωνήσω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να προωθήσουμε την έρευνα, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μην δώσουμε ειδική υποστήριξη μόνο σε δύο Ινστιτούτα που ξεχωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προτείνω έξι Ινστιτούτα όπως ε, ισχύει και στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Και έτσι θα μπορέσουμε να υποφεληθούμε από την προστιθέμενη αξία όλων αυτών των Ινστιτούτων ε, και όλη την ποικιλία που προσφέρουν. Πιστεύω επίσης ότι η δική μας Επιτροπή θα έπρεπε να επικεντρωθεί στους νέους που δεν έχουν πολλές δυνατότητες στη διάθεσή τους και είναι σημαντικό να λέμε ότι πώς ε, θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε την απασχόληση των ε, ατόμων που είναι κοινωνικό σε μειονεκτική θέση, των ατόμων με αναπηρίες. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτοί οι άνθρωποι να εκπαιδεύονται ώστε να μπορούν στη συνέχεια να εργαστούν και να ενσωματωθούν στην κοινωνία. Ευχαρίστω να ακούσω τις προτάσεις των συναδέλφων και αναμένω εναγωνίως την επικοδομητική μας συνεργασία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 Äh, hier äh, an die Arbeit geht. Und ich unterstütze das äh, vollinhaltlich und bemühe mich dort sicher, meinen Beitrag zu leisten. Danke. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο. Καστέλο. Κοστέλο. Συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και εγώ την εισηγήτρια για την εξαιρετική τη έκθεση. Εγώ συμφωνώ με όλη μου την καρδιά με τις συστάσεις της ε, εισηγήτριας. Ε, να πω ότι με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό το θέμα προσωπικά γιατί έχω εργαστεί για 10 χρόνια στην αρμόδια εθνική μας υπηρεσία που ε, διχειριζόταν τα προγράμματα κομίνιους και με ιδιαίτερα ενδιαφέρον τα θέματα σχετικά με τα προγράμματα διαβιομάθηση. Παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον όσα υπόθεσαν για την εκπαίδευση ενηλίκων και τη διαβιομάθηση. Είναι πραγματικά κρίμα ότι μόλις 2% ε, του προπολογισμού ε, θα διατεθεί σε αυτό. Ζητώ συγγνώμη για το κινητό μου. Αυτά είναι τα βασικά που θα ήθελα να πω σε αυτή τη φάση. Να πω ότι χαιρετίζω την πρόταση το πρόγραμμα αυτό είναι απαραίτητο, υποφελές και υποστηρίζουμε και αυτή την ιδέα για ένα ξεχωριστό πρόγραμμα για την νεολαία. Ότι είναι λάθο να τα βάζουμε όλα μαζί και ναι, είναι και ενιαίο ο χρηματοδοτικό φάκελο, θεωρούμε. Επίση, είναι ένα θέμα ε, επικουρικότητα και εθνικέ αρχέ θα πρέπει να αναλαμβάνουν στερή δράση τομέα αυτό. Αυτά προ το παρόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι υπάρχει εκπρόσωπο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλετε να πάρετε το λόγο? Πριν σα δώσω το λόγο, θα ήθελα να σας ε, ζητήσω το εξής. Δεν είμαι πάντοτε ο δικηγόρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά αν θέλουμε να μην υπάρχει κατακαιρματισμός και να δώσουμε κάποια ορατότητα στο πρόγραμμα αυτό, ε, το οποίο είναι μία από τις ε, καλές πολιτικές ε, που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, έχει μεγάλη επιτυχία και ιδιαίτερη ταυτότητα. Νομίζω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ως σημείο αφετηρία σε αυτό ακριβώς το σημείο. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος ο έρασμος να προαγάγουμε την ευρωπαϊκή δράση είχα την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το πρόγραμμα αυτό ήθελε ακριβώς να αυξήσει την ορατότητα, την ε, ε, εμβέλεια που θα κάλυπτε ε, το πρόγραμμα αυτό. Έχω την εντύπωση ότι όλοι όσοι έχουν ζήσει τα προηγούμενα προγράμματα δεν συμφωνούν ιδιαίτερα και νομίζω ότι θα έπρεπε ίσως να δείξουμε λίγο πιο έτσι, δυναμική ευφυΐα, για να το πω έτσι, σε ένα σημείο, σε μια χρονική στιγμή πολύ σημαντική. Συμφωνώ βέβαια ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στους νέους που βρίσκονται ανάμεσα στην, στον εκπαιδευτικό και τον επαγγελματικό βίο αλλά δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι το πρόγραμμα το οποίο συζητούμε τώρα είναι ο καλύτερος τρόπος να το κάνουμε αυτό. Η Επίτροπος Βασιλείου ήθελε ακριβώς να δείξει ότι είναι υπέρμαχος αυτής της ε, ιδέας του ε, προγράμματος έρασμος για όλους ε, Κρίμα που καμία από τις ε, ημερομηνίες που τις ε, ζητήσαμε να παραστεί δεν μπόρεσε να ε, είναι εδώ. Εγώ ευχαρίστω βέβαια να έχω μια ανταλλαγή απόψεων μαζί της αν το επιθυμεί στο περιθώριο των συνεδριάσεων του Στρασβούργου ενδεχομένω. Θα είναι χρήσιμο. Θα δούμε τώρα κατά πόσο θα γίνει. Συγγνώμη που πλατείασα λιγάκι αλλά θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια υποστήριξη. Χαιρόμεθα ιδιαίτερα γιατί αυτή η συζήτηση γίνεται εδώ στη δική σα επιτροπή. Καθώ και εμεί συμφωνούμε ότι συμβάλλετε τα μάλα στην όλη συζήτηση για το πράγμα για την εκπαίδευση, όπω πολύ ορθά είπατε, στόχο να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην ε, παιδεία και την ε, απασχόληση. Αν μου επιτρέπετε να κάνω για κάποια σχόλια για όσα ακούστηκαν. Πρώτα απ' όλα, ε, η ολοκληρωμένη προσέγγιση και το σκεπτικό πίσω από την πρότασή μας. Προσπαθήσαμε, αν θέλετε, να κάνουμε κάποιες αλλαγές σε σχέση με τα κείμενα προγράμματος, ώστε να κινηθούμε σε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Πιστεύουμε ότι όλα τα θέματα που άπτονται της παιδείας και της νεολαίας θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ολιστικά χωρίς κατακρεματισμό. Δείτε για παράδειγμα την πρώτη κατάληψη του σχολείου, είναι ένα θέμα που αφορά το σχολείο, την παιδεία, αλλά αφορά και την επαγγελματική ε, εκπαίδευση, κατάρτιση και την εκπαίδευση. πρέπει λοιπόν να βρούμε λύσεις που να καλύπτουν όλα τα παιδεία το ίδιο και για την ενσωμάτωση των μειονεκτικών ομάδων. Είναι κάτι που αφορά όλους τους τομείς της παιδείας. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε τη συνεργασία μεταξύ όλων, μεταξύ ε, της εκπαίδευσης, της νεολαίας κτλ. Το ίδιο και για τη διαφορετικότητα μέσα στη σχολική αίθουσα. Δηλαδή, πράγματα που αφορούν μεν τα σχολεία αλλά και την επαγγελματική κατάρτιση, την ανώτερη εκπαίδευση κτλ. Άρα αυτή είναι η βασική μας ιδέα πίσω από την πρόταση. Να προσπαθήσουμε να δούμε τα πράγματα μέσα από μια ολιστική προσέγγιση που πάντοτε έχει ως γνώμονα τη διαβίου μάθηση. Και έτσι πιστεύουμε ότι οι Έλληνες ενδιαφερόμενοι και οι ετούντες μπορούν ε, να βρουν μια λύση εκμεταλλευόμενοι αν θέλετε αυτή την ε, προσέγγιση τη σφαιρική. Τώρα, για τα ποσά. Θέλω να, να κάνω κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με το τι εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε. Ε, στην ανακοίνωση που συναδεύει την νομική βάση, να θέσουμε δηλαδή κάποια ποσοστά που θα εγγυόμαστε σε κάθε κλάδο, ακριβώς να μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλοι θα κερδίσουν από αυτή την ενσωμάτωση. Από το 2% ε, και το 7% για την εγκατάλειψη σχολείου δεν είναι τα ποσοστά που θέλουμε να πάνε κατακαιρματισμένα, αλλά είναι τα ποσοστά που τουλάχιστον θα συμβάλλουν στην περίοδο 2014-2020 αυτοί οι τομεί να λάβουν τουλάχιστον την, το ίδιο επίπεδο χρηματοδότηση όπω την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Δηλαδή, η ιδέα ποια είναι. Να αγγιθούμε το ίδιο επίπεδο χρηματοδότηση χρησιμοποιώντας δηλαδή από κοινού την αύξηση του προπολογισμού, δίνοντας πιο πολλά κονδύλια σε όλους τους επιμέρους τομείς. Τρίτο σημείο που θέλω να φέρω είναι η διεθνής διάσταση, κάτι που ανέφερε και η εισηγήτρια. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι αυτή είναι η πρόταση Ερασμός ε, για όλους. Έχει τις απαρχές 7 χωριστά προγράμματα, 5 εκ των οποίων αφορούν την διεθνή διάσταση της εκπαίδευσης, Ερασμούς Μούντους, Τέμπους, Αλφα κτλ. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα προγράμματα που ήδη τρέχουν τώρα, ακριβώς που αφορούν τη διεθνή διάσταση και ενσωματώνονται εδώ. Και ειδικά βεβαίως ξεχωρίζει εδώ η νοτρική εκπαίδευση εν προκειμένου τα ιδρύματα ανώτερη εκπαίδευση βεβαίω κινούνται σε ένα παγκοσμιοποιημένο, αν θέλετε, ε, πεδίο, κάτι που δεν ισχύει για όλου του άλλους τομείς και γι' αυτό και η χρηματοδότηση για τέτοιου είδου δραστηριότητε δεν προέρχεται από τον έρασμο για όλους, αλλά από άλλα εργαλεία, όπως το εργαλείο για την αναπτυσιακή συνεργασία και εκεί πραγματικά αναφέρουμε ρητά ότι κάποια κονδύλια θα μεταφερθούν ειδικά για το τον έρασμο για τη συνεργασία στην ανώτερη εκπαίδευση. Και γι' αυτό έχουμε και την κατάλληλη νομική βάση. Και δύο ακόμη σημεία. Πρώτα απ' όλα για τι δράσει Jean Monnet. Τα δύο θεσμικά όργανα που αναφέρονται στην νομική βάση, και εδώ έχουμε την πρόταση τη εισηγήτρια να προσθέσουμε και άλλα. Υπάρχει λόγος στον οποίο εμεί δεν κάναμε μία πρόταση για έξι προτινόμενα ιδρύματα. Αυτό που θέλουμε να ε, ε, προάγουμε είναι η αριστεία στην ε, εκπαίδευση, αλλά θεωρούμε ότι υπάρχουν και πολλά ευρωπαϊκά ιδρύματα που θα μπορούσαν να λάβουν αυτή τη χρηματοδότηση επάξια. Θα το δείτε και ιστορικά. Είναι πάρα πολλά τέτοια τα ιδρύματα που δίνουν πολύ ψηλέ υπηρεσίες υψηλή ποιότητας. Με τον ανταγωνισμό, την ευγενή άμυλα αν θέλετε, και την υποβολή έκφραση ενδιαφέροντος για κάθε project, για μακροχρόνια χρηματοδότηση, είναι καλύτερο παρά να περιορίσουμε και να ορίσουμε συγκεκριμένα ιδρύματα σε μια νομική βάση. Έτσι θα εξαλειφθεί το στοιχείο της άμυλας. Και τελευταίο σημείο που συνδέεται και με τα εισαγωγικά σχόλια της Προέδρου. Ποια είναι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό σε σχέση με το παρελθόν. Αναγνωρίζουμε ότι παρά το συνολικό ποσό που θα αποσπάσουμε, ουσιαστικά, αντικειμενικά μιλάμε για ένα πολύ χαμηλό ποσό. Άρα λοιπόν είναι προς το όλων να δοθούν αυτά τα χρήματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με αυτή τη νομική βάση λοιπόν αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να εστιάσουμε τη χρηματοδότηση στους τομείς εκείνους όπου θα δώσουν την μεγαλύτερη και καλύτερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Γι' αυτό έχουμε κάνει αυτές τις επιλογές. Πρόθεση της ε, κινητικότητας των εκπαιδευτών, των, ε, του εκπαιδευτικού προσωπικού, διότι όταν πηγαίνουν στο εξωτερικό ε, και μαθαίνουν νέες μεθόδους, βλέπουν άλλα πράγματα, η εκπαιδευτική αυτό είναι προς όφελος όλων των ε, μαθητών, των ενήλικων μαθητών. Θεωρούμε λοιπόν ότι η ε, επένδυση, αν θέλετε, η χρηματοδότηση κινητικότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι προς όφελος όλων. Όπως επίσης αυτό ενισχύει και τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ενδρυμάτων. Ελπίζω τουλάχιστον να πάτε σε κάποια από τα σημεία που σας απασχολούν και προσβλέπουμε και εμείς σε περαιτέρω συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λύση συγκήτρια. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπέκερ και την κυρία Κοστέλο Προσβλέπω σε στενή συνεργασία μεταξύ μας. Αν έχετε προτάσεις, ε, τροπολογίες ε, για την γνωμοδότηση την οποία συντάσω, ε, Ευχαριστώ να τις ακούσω. Όσον αφορά στις απαντήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ και σας ευχαριστώ πολύ για την άποψή σας. Δεν συμφωνώ όμως με όλα όσα είπατε. Μιλήσατε για την διάσταση της διεθνούς συνεργασίας και είπατε ότι τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης ε, όπως αναφέρεται και στον κανονισμό, έχουν επαρκή χρηματοδότηση. Από την άλλη λέτε όμως ότι πρέπει να υπάρξουν και καινοτόμοι δράσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν για ποιο λόγο δεν μπορεί αυτή η πτυχή να συμπεριληφθεί στη διεθνή διάσταση. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν πραγματικά πολύ εποφελές και νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε μια λύση σε σχέση με αυτό όσον αφορά κάποια, ε, κάποιες ποσοστιαίες μονάδες που αναφέρατε. Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα προγράμματα δεν πρέπει να λάβουν μικρότερη χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη ε, για την, για όλη, όλα τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης, γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι αυτό που παράγει ε, δημόσια ε, κοινοφελή αγαθά. Αν θέλουμε λοιπόν περισσότερη χρηματοδότηση, η χρηματοδότηση αυτή πρέπει να κατανεμηθεί σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εγώ όταν συνέταξα τη γνωμοδότησή μου δεν ήθελα να αντιπαραβάλω τον έναν εκπαιδευτικό τομέα με τον άλλον. Απλώς δίδεται προτεραιότητα στην επόμενη προγραμματική περίοδο στην ανώτερη εκπαίδευση. Μην όμως ξεχάσετε τους υπόλοιπους τομείς. Αυτό είναι το μόνο που ζητώ. Ας δούμε την πραγματική κατάσταση και τις ανάγκες των πολιτών μας. Και βεβαίως οι ανταλλαγές αυτές ε, σημαίνουν προστιθέμενη αξία και ωφέλη στον τομέα της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω λοιπόν να καταλήξουμε σε μια συμφωνία μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι θα θέλαμε να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο Βασιλείου, αλλά δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν. Εν πάση περιπτώσει, εμείς προτείναμε κάποιες ημερομηνίε. Λοιπόν, Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 27 Αυγούστου στις 2 ε, το απόγευμα, 17 και 18 Σεπτεμβρίου θα τις εξετάσουμε, κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει να εξετάσουμε τις συμβιβαστικές 8 Οκτωβρίου και να ψηφίσουμε την επομένη 9 Οκτωβρίου. Η Επιτροπή ε, Πολιτισμού θα ψηφίσει τις 6 Νοεμβρίου. Ολοκληρώσαμε και το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης και φτάνουμε στο τελευταίο μας σημείο πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές που είναι το σημείο 22 εξέταση των τροπολογιών στην έκθεση της ε, κυρίας Μπίργκιτ Σίπελ γνωμοδότηση για την επί της Επιτροπή ΙΜΚΟ σε σχέση με την σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Επειδή η κυρία Σίπελ όμως δεν είναι εδώ, η κυρία Ρέγνερ θα ε, την ε, αντικαταστήσει. Της δίνω το λόγο.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 Θα ήθελα απλώ να υπενθυμίσω ότι αν υπάρχουν τροπολογίε οι οποίε δεν αφορούν ε, τι αρμοδιότητε τη Επιτροπή ε, Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων, θεωρούνται μη παραδεκτέ. Οπότε σα το λέω αυτό γιατί έτσι θα διευκολυνθεί το έργο τη εισηγήτρια. Θα το δούμε τέλο πάντων με την εισηγήτρια και με τους ε, υπολείπους συναδέλφους ε, γιατί ούτως ή άλλως μπορούν οι εισηγητές συνήθως να ε, εισαγάγουν μία πτυχή κοινωνική ώστε να μπορούν να θεωρηθούν παραδεκτές τροπολογίες. Η κυρία Εσάγια. Ευχαριστώ. Ε, πρόεδρε, θα χρήσω στη μετρική μου γλώσσα, στα φιλανδικά, και θα πω ότι ευχαριστώ θερμά την εισηγητρία και την καλή προσπάθεια που έκανε και για το γεγονός ότι ήδη προχωρήσαμε στην κατάρτιση των συμβαστικών προτάσεων ήδη από το Στρασβούργο. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτούς τους ρυθμούς για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε τελικά τις θέσεις του συνομοθήτη σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις. Είναι πολύ σημαντικό ε, να καταλήξουμε σε ένα κείμενο απλό, εύληπτο, κάτι που είπα ήδη και στη συνάντησή μας στο Στρασβούργο. Είναι πολλά τα μείζωνα ζητήματα που αφορούν ε, την προστασία και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Δεν μπορούμε, πιστεύω, να ορίσουμε χωριστά τους όρους και τις ρήτρες που θα περιέχουν αυτές οι συμβάσεις χωρίς να λάβουμε υπόψη τα δικαιώματα των εργαζομένων, ιδίως για τις τροπολογίες Θέλω να αναφερθώ στις δικές μου τροπολογίες που αφορούν ένα σύστημα παροχής υπηρεσιών μέσω voucher. Είναι κάτι που χρησιμοποιούμε πολύ συχνά, είναι πολύ διαδεδομένο στις σκανδιναβικές χώρες για την καλύτερη οργάνωση της παροχής υπηρεσιών και φαίνεται ότι είναι κάτι που αποδίδει. Έχουμε παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με αυτόν τον τρόπο επίσης ε, με έναν τρόπο διασφαλίσει και ε, το υψηλό επίπεδο των παρόχων υπηρεσιών. Η χρήση λοιπόν αυτών των voucher παροχής υπηρεσιών είναι μια εγγύηση ποιότητας τροποντινά. Αυτά τα voucher επίσης θέλω να πω επιτρέπουν και στις μικρές επιχειρήσεις, ακόμη και τις ατομικές επιχειρήσεις, να συμμετάσχουν σε τέτοια εγχειρήματα. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα ήταν καλό να υπάρξει και να εισαχθεί αυτή η ιδέα ε, στην ε, έκθεση Πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει σε ένα καλύτερο σύστημα σε όλη την Ευρώπη. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο άρθρο 11 ετάχη που αφορά τις διακυβερνητικές σχέσεις. σχετικά με, τα, με το ίδιο ιδιοκτησίας αυτές τις εταιρείες. έχουμε γίνει μάρτυρες κάποιων αρνητικών εκπλήξεων στο παρελθόν σχετικά με τη μορφή και το καθεστώς που έχουν αρχικά τέτοιες επιχειρήσεις και τι τελικά, ε, σε τι τελικά εξελίσσονται. Δηλαδή πόσο μερίδιο, αν θέλετε, αυτών επιχειρήσεων μπορεί να πάει σε ιδιωτικά χέρια. Είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να αφήσουμε στην άκρη. Επίσης, ένα άλλο σημείο της πρότασης σχετικά με τη δικαστική εποπτεία, με την έλλειψη πρόβλεψης στην πρόταση για επιβολή κυρώσεων Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που λείπει, αλλά και να αναφερθώ και στο άρθρο 7.3, το οποίο θεωρώ ότι είναι και αρκετά προβληματικό και δύσκολα εφαρμόσιμο. Ούτως ή άλλως, όλα τα κράτη-μέλη έχουν τη δική τους εθνική νομοθεσία περί ε, συμβάσεων που ρυθμίζουν τις πιο πολλές πτυχές ε, των ε, θεμάτων που ήδη θίγει και αυτή η γνωμοδότηση. Πολλοί ε, αναφέρονται βεβαίως και στη σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. και αν έχω καταλάβει καλά και το Συμβούλιο αντιμετωπίζει αρκετές διαφωνίες στο ιστορικό του σχετικά με τη σύμβαση της Διεθνού Οργάνωση Εργασία κατά όσο να συμπεριληφθεί ή όχι. Αυτό αφορά το άρθρο 23 της ε, πρώτη οδηγία. Για τα άρθρα 25 και 26 υπέβαλα και εκεί κάποιες τροπολογίες για καταληκτικές προθεσμίες, ώστε να διευκολύνουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έπειτα για τα πρότυπα και τις επισημάνσεις ε, το κόστος του κύκλου ζωής και κάποιους άλλους ορισμούς, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ξέρετε, υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί και θα πρέπει η μέθοδη υπολογισμού να είναι διαφανής και προσβάσιμη σε όλους, ώστε να μην είναι εύκολες οι αθέμετες πρακτικές. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Κύριε Μπουλό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια ε, για τη δουλειά της μέσω της κυρίας Νέγνερ, αλλά θα ήθελα να πω επίσης ε, ότι μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον για μένα, ενδιαφέρουσα για μένα αυτή η έκθεση σε σχέση με την εισαγωγή ε, κοινωνικών προτύπων στην σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερα στο βαθμό που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε τις, ε, τα ελάχιστα που πρέπει να υπάρχουν ώστε το αντικείμενο της ε, σύμβασης να είναι βέβαια σχετικό. Νομίζω όμως ότι από την άλλη πρέπει να μπορούμε ως επιπλέον παράγοντα στο, στην ε, ανάθεση μιας σύμβασης όχι να είναι μόνος ένα, ένας απαρέγκλητος παράγοντας, αλλά ε, να αναφέρονται επαρκώ κοινωνικοί, τα κοινωνικά πρότυπα, πρότυπα, όπως το αναφέρει η Διεθνή, Οργάνωση Εργασίας, για παράδειγμα, υπάρχει το θέμα του προσανατολισμού ε, της Δημόσιας Σύμβασης. Ε, κατά τη γνώμη μας δεν είναι παρκές αυτό. Πρέπει να πάμε λίγο ακόμα, λίγο ακόμη παραπέρα, ώστε να μπορούν να θέτουν ε, σημαντικούς κανόνες κοινωνικής αλληλεγγύης, να, να είναι κάτι το οποίο θα θέτουν στο οποίο θα δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα οι επιχειρήσεις, γιατί όχι να μην υπάρχει και μία σήμανση σε σχέση με το θέμα αυτό. Να μπορούμε δηλαδή να τονίσουμε, να δείξουμε κάποιες επιχειρήσεις ε, ως επιχειρήσεις που ε, είναι πιο κοινωνικές. Νομίζω ότι αυτός ο παράγων ανάπτυξης επιτρέπει μια κάποια σύγκληση, δηλαδή ε, μία ε, σύγκληση στο πλαίσιο μίας όλο και πιο ενιαίας αγοράς. Εγώ θα προτείνω τροπολογίες που πηγαίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Σκοπό έχουν να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στην εισαγωγή των κοινωνικών προτύπων. Υπάρχουν βέβαια και κάποια ζητήματα στο θέμα της υπεργολαβίας, ε, ε, στην ανάλυση των κριτηρίων των κοινωνικών, ε, αν πηγαίνουν πέρα από τα κριτήρια τα βασικά και τα υποχρεωτικά. Ποιο τα ορίζει, ποιο τα επιβλέπει, ποιο τα πιστοποιεί. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα συνεπώ που πρέπει να τεθούν για το θέμα αυτό, αλλά ε, συμφωνώ απολύτως ε, ε, με την εισηγήτρια. Μπορούμε να συνεργαστούμε και για συμβιβιστικέ τροπολογίες. Είμαστε νομίζω σε μία οδό σύγκλησης μεταξύ των πολιτικών μας ομάδων. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ρέγνερ, θέλετε να ξαναπάρετε το λόγο. Όχι, υπόθηκαν όλα. Κύριε Σέρκα, θέλετε να πάρετε το λόγο. Έχετε το λόγο. Eh, Όχι, Πρόεδρε, μόνο να επισημάνω την τεράστια σημασία που δίνουμε εν προκειμένου σε αυτό το θέμα και το πώς η φωνή της Επιτροπής Απασχόλησης θα πρέπει να εισακουστεί. Έχουμε να κάνουμε με έναν τομέα με πολύ ψηλό όγκο ποσών που θα κινούνται και θα πρέπει να υπάρξει και και κοινωνική διάσταση, αν θέλετε, και στη δημόσια που θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τον τελευταίο ομιλητή. Ελπίζω να μην έχουμε την εμπειρία που είχαμε στην προηγούμενη, σε μια προηγούμενη έκθεση νομίζω της κυρίας Ρούλε στην Ολομέλεια, η άποψη της Επιτροπής μας δεν ήταν καθόλου θετική συνεισφορά. Και το λέω αυτό όχι ως πρόεδρος της Επιτροπής, αλλά είναι ένα προσωπικό σχόλιο. Τέλο πάντων, δεν μου άρεσε ιδιαίτερα η τοποθέτηση τη Επιτροπή μα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εφόσον υπάρχει ένα πνεύμα συμβιβασμού, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να είμαστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω τη οποία θα μπορέσουν, θα, μπορέσουν οι, κοινωνικές, οι δημόσιε συμβάσει να συμπεριλάβουν αυτή τη διάσταση την κοινωνική να μην ε, αφορά μόνο την ε, ε, μειοδοτούσα προσφορά, να μην υπάρχει μόνο το κριτήριο της μειοδοτούσας προσφοράς. Θα ήθελα να υπενθυμίσω το χρονοδιάγραμμα, το οποίο το ανέφερε ούτως ή άλλως ε, και η ε, αντικαταστάτρια της εισηγήτριας. 17 Σεπτεμβρίου θα εξετάσουμε τις συμβαστικέ τροπολογίες, να τις εγκρίνουμε 18, ε, συγγνώμη. Η ΙΜΚΟ ψηφίζει στις 10 Οκτωβρίου για την έκθεση του συναδέλφου Μάρκ Ταραμπέλα ολοκληρώσαμε και το ε, σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχει τίποτε υπό τα διάφορα, σας δίνω ραντεβού για τις 6 Σεπτεμβρίου και σας εύχομαι πολύ καλές διακοπές. Γεια σας.